Ε, start Να ξεκινήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί νομίζω ότι είχε υπάρξει ένα μήνυμα για μια ψηφοφορία που θα γίνει νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί, αλλά δεν θα υπάρξει πρόορη ψηφοφορία. Ε, δεν ξέρω αν πήρατε το email, θα σας εξηγήσω. Θα ψηφίσουμε στις 9.30, αλλά όχι πριν εντάξει. Οπότε καθίστε με την ησυχία σας. Δεν θα ψηφίσουμε στις 9. Μην ανησυχείτε λοιπόν. Οπότε να ξεκινήσουμε. Έγκριση της ημερής σε διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνεται. Δεν έχω ανακοινώσει. Τα πρακτικά της συνεδρίας 18 Οκτωβρίου, 19 Νοεμβρίου, 24 Ιανουαρίου, 4 Φεβρουαρίου αν έχετε αντιρρήσεις εγκρίνονται. Και περνάμε τώρα στο πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη. Ο κύριος Βόμποντα δεν θα έρθει, δεν είναι σε θέση. Εγώ θα το παρουσιάσω λοιπόν. Όπως ξέρετε, είναι το πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη. Πήγα σε έναν από τους τριμερείς ε, διαλόγους τουλάχιστον. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν και το προσωπικό. Εργάστηκαν πολύ σκληρά για το πρόγραμμα αυτό και κατέληξε επιτυχώς. Όπως ξέρετε, προσωρινή συμφωνία επετεύχθη μετά τον πολιτικό τριμερή διάλογο της 5ης Μαρτίου. Το θέμα αντιμετωπίζεται με βάση το, κανόνα, το άρθρο 55. Ο κύριος Βόμποντα θα μας είχε ενημερώσει, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί. Μετά λοιπόν τις περαιτέρω τεχνικές συζητήσεις, τα επόμενα βήματα για το πρόγραμμα για το δικαιοσύνη, θα είναι η ενημέρωση από του δύο συνεισηγητέ για την κατάσταση πραγμάτων όσο αφορά τι διαπραγματεύσεις. Αυτό βεβαίως ε, δεν δημιουργεί προβλήματα. Λοιπόν, ας έχουμε αυτή την ενημέρωση. Έχουμε τον ε, ε, κύριο Βάιντεν Χόλτσα και την κυρία Χάουταλα. Ποιος θα πάρει πρώτο το λόγο? Ο κύριος Βάιντεν Χόλτσα. Ναι, σύντομα. Σημειώθηκε ουσιώδης πρόοδος. Έγιναν ε, ουσιώδεις αλλαγές. Οι διαπραγματεύσεις πήγαν πολύ καλά και γρήγορα. Καταλήξαμε σε μερική συμφωνία. Λύσαμε και τα προβλήματα για το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και τις αξίες. Τώρα βέβαια δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει η θέση του Συμβουλίου. Καλό θα ήταν να διευκρινιστεί πόσο ταχύτερα γίνεται. γιατί θα ήταν κρίμα να πάει χαμένη όλη αυτή η δουλειά λόγω των αβεβαιοτήτων. Η Χάιντι ξέρει πιο πολλά για το διαδικαστικό. Η διάσκεψη των Προέδρων ε, συνεδριάζει τώρα, οπότε ίσως να διευκρινιστεί η κατάσταση μετά τη συνεδρίασή της και μετά να ψηφίσουμε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι συζητάνε. Ευχαριστώ, Τζο. Αλλά για να ελέγξω αυτή η επιστολή του Συμβουλίου δεν ε, θίγει τις προθεσμίες για να έχουμε τροπολογίες ε, και κείμενα για την ε, Ολομέλεια του Απριλίου, τη δεύτερη. Η Χάιντι. Οι συνεισηγητές είναι ικανοποιημένοι με το περιεχόμενο αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι με ε, την πλευρά που σχετίζεται με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο όπου δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η επιστολή αυτή έχει ημερομηνία 19 Μαρτίου, τη λάβαμε στις 20 και λέει ότι είμαστε πεπισμένοι ότι αν υπάρχει ένας βαθμός ε, βεβαιότητα για τα επόμενα πολιτή προγράμματα θα δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τα μέσα από την αρχή του νέου πολιτού πλαισίου. Το Συμβούλιο περιμένει ότι οι διαπραγματεύσει με το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ξεκινήσουν όσο να το πιο σύντομα για να ολοκληρωθούν με βάση την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί και που αναφέρεται στην κοινή κατανόηση χωρίς όμως ε, αυτό να προδικάζει της ε, την κατάληξη των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 21-27. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι το Συμβούλιο δεν θα ακυρώσει εντελώς την μερική συμφωνία που έχουμε του περιεχομένου. Όπως είπε και ο Τζο, είναι λυπηρό που κάνουμε τη, στιγμή, τη συζήτηση μας αυτή τη στιγμή που η διάσκεψη των Προέδρων συζητάει πώς θα αντιδράσει συνολικά το Κοινοβούλιο στην επιστολή του Συμβουλίου. Νομίζουμε ότι σε αυτή τη συγκυρία δεν θα είχε έννοια να ψηφίσουμε. Θα μπορούσαμε όμω να ψηφίσουμε στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια αργότερα. Γιατί δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει η διάσκεψη των Προέδρων. για αυτό το δίλημα. Έτσι είναι τα πράγματα. Τζο, θες να προσθέσεις, όχι. Ε, ωραία. Λοιπόν. Καταρχάς σας ευχαριστώ και πάλι για την εργασία που κάνατε, γιατί παρακολούθησα τους τριμερείς διαλόγους εν μέρη. Ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ για την ενημέρωση για την επιστολή του Συμβουλίου. Προφανώς είναι ένα θέμα που θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε. Αλλά φυσικά θα συνεχίσουμε με βάση το πρόγραμμα εργασιών μας μέχρι τη δεύτερη ολομέλη του Απριλίου, αλλά θα δούμε και πώ θα αποτιμήσει η διάσκεψη των Προέδρων την ε, επιστολή του Συμβουλίου. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι του συζητητές και όλου όσου ε, συμμετείχαν ε, στην εργασία για το θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ. Και βεβαίω θα ψηφίσουμε στη δεύτερη του Απριλίου, στη δεύτερη ολομέλη του Απριλίου, όταν αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε, σημείο 2. Λοιπόν, αυτή ήταν μια κοινή συνεδρίαση Λίμπε και Τζούρι. Λυπάμαι που είμαι μόνο εγώ, αλλά δυστυχώς ο κύριος Βόμποντα ε, δεν μπορεί να παρευρεθεί. Και ζητά συγγνώμη. Είχε άλλες υποχρεώσεις. Λοιπόν, να, να συνεχίσουμε τώρα με τη συνεδρίαση της Λίμπε. Λοιπόν, έγκριση των πρακτικών. Λοιπόν, έχουμε τη στάδια αλλαγές στο σχέδιο μέσα Το σημείο 8 η ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης για τη διάδοση ε, διαδικτυακού τρομοκρατικού περιεχομένου θα γίνει στη συνεδρίαση μας 1η και 2η Απριλίου, στο σημείο 10. Ψήφος για την προσωρινή συμφωνία μετά από διοργανικές ε, διαπραγματεύσεις για το κατάλογο των τριών, τρίτων χωρών των οποίων ε, οι υπήκοοι πρέπει να έχουν προξενικές θεωρήσεις και αυτό έχει αναβληθεί. Έχουμε ένα νέο α, το, η, ψήφιση, το, η ψηφοφορία για μια Ευρώπη που προστατεύει, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να επεκταθούν οι δραστηριότητες του εισαγγελέα στις διαμεθοριακές ε, τρομοκρατικές ενέργειες στις 9.30 15. Ε, τα θέματα της ΛΥΜΠΕ για το πολιτές πλαίσιο 2021-2027 θα γίνει σε 9.35 αντί για τις 11.50 Σημεία 18 και 20. Η παρουσίαση των σχεδίων εκθέσεων για τα συμπεράσματα των συμφωνιών μεταξύ με της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, της Σερβίας, ε, του Μαυροβουνίου, της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης και η δράση από την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή αναβάλλεται και σημείο 17 ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις για την ε, Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Εκτοφυλακή θα γίνει στις 15 και 15 και 14.45. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, εγκρίνεται αυτή η μερίσια διάταξη. Οπότε, γλώσσες. Διερμηνία σε όλες τις γλώσσες εκτός από δανέζικα, κροατικά, ε, μαλτέζικα και γοηδελικά. Ε, αποφάσεις των συντονιστών 2.5, ε, άρθρο 205. Εισηγητές δηλαδή. Ποιοι ορίστηκαν ως εισηγητές. Η Ρομπέρτα Μετσόλα από το ΕΛΚΑ. Γεια σου Ρομπέρτα. Είναι μεγάλο δωμάτιο και είμαι εδώ, διαβάζω εχόμενα στα χαρτιά μου. Γιατί φοβάμαι αυτό που θα δω. Μήπω συμβεί τίποτα. Αλλά καλώ ήρθες. Ρομπέρτα λοιπόν, είσαι εισηγήτρια για τα εξή θέματα. Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Λίχτενστάιν για, την... Ε, για μια σειρά πράγματα. Κατά πολέμης τρομοκρατία, διαμεθοριακό έγκλημα κτλ. Είναι μια απόφαση πλαίσιο. Επίση, συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση και Σουηδική, ε, ε, Ελβετική συγγνώμη Ομοσπονδία για διάφορα θέματα επίση Λοιπόν, εγκρίνεται αυτές τις συστάσεις. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ε, κατεξοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις. Λοιπόν, θα τα πω στα γρήγορα. Υπομονή. Στις 12 ε, Μαρτίου το Κοινοβούλιο έλαβε τέσσερα ε, σχέδια εφαρμοστικών πράξεων. Ο κανονισμός 515-2014 ε, ε, για το αιτία. οι τέσσερις ε, εφαρμοστικέ πράξεις που αφορούν το αιτία, Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για, την, στάνταρ, για το στάνταρ έντυπο για την ακύρωση του κανονισμού 2018-1240 ένα, ένα σχέδιο απόφασης για τις προϋποθέσεις προσωπικών δεδομένων που θα πρέπει να μπουν στο έντυπο και για τις παραμέτρους για την εξακρίβωση που πρέπει να γίνει για να, διαμορφωθεί, για να διαπιστωθεί αν είναι πλήρης η αίτηση. Σχέδιο εφαρμοστικής απόφασης για τη διατήρηση και πρόσβαση στα αρχεία του αιτίας ε, με βάση το αρθρο 933 73.3β του κανονισμού 2018-2040 και τέλος σχέδιο εφαρμοστικής απόφασης για τις τεχνικές λύσεις για να συνδέονται τα κεντρικά σημεία του ΕΤΙΑΣ με τα περιφερειακά σημεία και μια τεχνική λύση για να διακολυνθεί η συλλογή στοιχείων από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπόλ για να ε, ε, εκπονούνται στατιστικές για την πρόσβαση στα στοιχεία του ΕΤΙΑΣ για αστυνόμευση. Η λήψη αυτών των ε, εφαρμοστικών πράξεων ανακοινώθηκε μέσω της, του newsletter μας και υπάρχει εσωτερική προθεσμία για αντιρρήσει, Αν έχετε αντιρρήσει, παρακαλώ να ενημερώσετε τη γραμματεία μας πριν τι 26 Μαρτίου 12 το μεσημέρι. Στις 12 Μαρτίου το Κοινοβούλιο έλαβε αποφάσεις για εφαρμοστικέ πράξεις ε, παρόμοιε, οι οποίες αφορούσαν τον κανονισμό 2017-226 συγγνώμη 2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10 του Νοεμβρίου 2017 για ένα σύστημα εισόδου-εξόδου, το EES. Η εισαγωγή αυτή τη εφαρμοστική πράξη ε, απεστάλλει σε εσά μέσω του newsletter 15 Μαρτίου και πάλι υπήρξε εσωτερική προθεσμία. Υπήρξε λοιπόν μια εσωτερική προθεσμία για αντιρρήσει. Εάν ε, θέλετε να θέσετε αντιρρήσει, να ενημερώσετε την γραμματεία μα πριν τι 26 Μαρτίου 12 το μεσημέρι. Και θα ψηφίσουμε στι 9.30 σήμερα να έχετε τι ηλεκτρονικέ σας κάρτες. Και η έγκριση των πρακτικών, το συνέδριό είναι 7 Ιανουαρίου, 19 και 20 Νοεμβρίου πέρυσι, 5 Νοεμβρίου, 28 Ιουνίου, 25-26 Απριλίου, 12 Απριλίου, 9 Απριλίου, 19-20 Φεβρουαρίου, 20 Φεβρουαρίου και πάλι, 24-25 Ιανουαρίου. Λοιπόν, για όλα αυτά τα πρακτικά, αν δεν έχετε αντιρρήσει εγκρίνονται. Ωραία. Κάναμε τα 5, 6 και 7. Ο συγητής ο κύριος Κοράου δεν είναι εδώ. Η ε, κύριε Δία δεν έχετε πρόβλημα με τη διερμηνία. Όχι, α, ωραία. Εντάξει, ακούτε. Ο συγητής μα δεν είναι εδώ. Λοιπόν, συνάδελφοι. Δεν είναι εδώ ο κύριος Κοράου. Ψηφίζουμε στις 9.30. Λοιπόν, σύντομη διακοπή. Καφέ, χαλαρώστε. Θα ψηφίζαμε τώρα, αλλά... Αλλά μ, δεν είμαστε και τόσο πολλοί. Καλά δεν είναι και ψηφοφορία που θα μας πάρει πολύ ώρα. Sorry for the delay, colleagues. Uh, Mr. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αν έρθει ο κύριο Κοράο, θα του δώσω τον λόγο. Ε, δεν θα καθυστερήσουμε. Αλλά αλλιώ σύντομο διάλειμμα. Και στις 9.30 ακριβώς θα αρχίσει η ψηφοφορία. Γιατί ξέρω ότι ορισμένοι να φύγουν, είναι πέντε πρωί. Yeah. Um, να περάσουμε στην ψηφοφορία, παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, ξεκινάμε με τη θέσπιση του προγράμματος Δικαιώματα και Αξίες. Μποντήλ Βολέρη, εισηγήτρια. Θα θέλατε το λόγο. Πολύ σύντομα να πω ότι ολοκληρώσαμε το έργο μας που ήταν άκρο δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την σημερινή ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Λάβαμε δε μία επιστολή από το Συμβούλιο την οποία είχαμε ζητήσει εμείς για να μας επιβεβαιώσουν ότι συμφωνούν με όλα όσα συμφωνήσαμε αμφότερες οι πλευρές. Λάβαμε αυτή την επιστολή. Βέβαια, υπάρχουν κάποια ζητήματα που εκκρεμούν ακόμη ό,τι είναι σε αγγείλες δηλαδή και τα λοιπά. Αυτά θα τα δούμε αργότερα. Ευχαριστώ πρόεδρος, ευχαριστώ Μποντήλ. Περνούμε στην ψηφοφορία, ηλεκτρονική νέα ψηφοφορία, το σύνολο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τόμας, Κρατάω την ψηφοφορία να καθίσει και εσύ να ψηφίσει. Παρακαλώ ψηφίστε συνάδελφοι. This is worth voting for. Okay, everyone's... Ψηφίσατε όλοι. Πέρασες τη ψηφοφορία 31 ψήφοι 3 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, την Ποντήλ. Επόμενη. Να σας διαβάσω μια σύντομη εισαγωγή τη διαδικασία για αυτό το σχέδιο ψηφίσματος της ΛΥΜΠΕ επειδή ήταν ε, κάπως ταχαία η διαδικασία δεξιγματικά να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την Ευρώπη που προστατεύει την πρωτοβουλία για την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Γραφείου Αγγελία ε, για να καλύπτονται και τα ε, τρομοκρατικά εγκλήματα. Από ό,τι ξέρετε, υπάρχει το μέρο ε, τη επέκταση ε, των αρμοδιοτήτων. Ο ΕΠΟ θα είναι υπεύθυνο για τα λεγόμενα δικήματα ΠΙΦ, κατά δηλαδή των χρηματοπιστωτικών σφαιρόντων τη Ένωση και τα συναφή με αυτά αδικήματα. Η δομή λοιπόν του Ευρωπαϊκή Αγγελία κατά πάσα πιθανότητα θα είναι επιχειρησιακή στα τέλη του 2020 ή στι αρχέ του 2021. Το συγκεκριμένο ψήφισμα ζητά, από, ζητά ενδεχόμενη δυνητική πάνω, παράταση ε, επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαίου Εισαγγελέα για να αντιμετωπίσει και τα διασυνοριακά τρομοκρατικά δικήματα. Αυτό είναι δυνατό δυνάμε το άρθρο 86 τη τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ενεκρίθη αρκετά αργά. Αυτό είναι σημαντικό για εμένα. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια, μπορώ να περάσω θες αμέσως στην ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα έχουμε την τροπολογία 1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και πηγαίνουμε στην τροπολογία 2, άρχεται η ψηφοφορία. Μάιτε. Δεν είσαι μαζί σου την κάρτα σου. Άρα θα καταγράφουν την ψήφο σου. Για να βάλω τα ακουστικά μου, παρακαλώ. Α, απλά λες τι ψηφίζεις, εντάξει. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και να καταγραφεί η ψήφος της ΜΑΙΤΕ. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Μάλλον άρχεται. Είναι ανοιχτή ψηφοφορία. Πέρας το όπως και προηγούμενη. Πηγαίνουμε στην τελική ψηφοφορία, ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 33 ψήφους υπέρ, 5 κατά, 2 αποχές και εδώ ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Uh, dear colleagues, um, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα επανέλθω στην ημερήσια διάταξη. Είναι πέμπτη πρωί και γνωρίζω ότι υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι οι οποίοι φεύγουν. Τέλο πάντων φύγετε, αλλά ησύχω ε, το επιθυμείτε για να περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, ε, το σημείο 15 που είναι το πολιετέ μεσονομικό πλαίσιο, παρουσίαση τη ε, τρέχουσα κατάσταση. Όποιοι θέλετε να ακούσετε, να ακούσετε παρακαλώ. Όποιοι θέλετε να αποχωρήσετε, αποχωρήστε. Σας κάνω λοιπόν μια επικαιροποίηση για τα θέματα που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο ως πρόεδρος ομάδας επαφής της ΛΥΠΗ για το ενδιάμεσο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 21-28 θα ήθελα να σας ενημερώσω για το πώς προχωρούμε με τα διάφορα τομεακά προγράμματα για τα οποία έχουμε αρμοδιότητα ως Επιτροπή. Πρόκειται συγκεκριμένα για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, για το Ταμείο Στερικής Ασφάλειας, ε, για το Ταμείο Διαχείρισης Συνόρων και Θεωρήσεων, το Ταμείο Περικλής, ε, το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων και Αξιών και το Πρόγραμμα Δικαιοσύνη. Ποια είναι η διαδικασία Όπω γνωρίζετε, αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων πω όλε οι εκθέσει που σχετίζονται με το πολιτέ μεσονομικό πλαίσιο πρέπει να έχουν κλείσει πριν τα τέλη τη θητεία, ε, στο πλαίσιο τη πρώτη ανάγνωση, έχοντα υπόψη ότι προ το παρόν μπορούν να συναφθούν με το Συμβούλιο μόνο μερικέ σύμφωνε. Στι περιπτώσει εκείνε όπου οι διαπραγματεύσει ε, με το Συμβούλιο έχουν ολοκληρωθεί, θα πρέπει να αποφασίσει η διαπραγματευτική ομάδα κατά πόσο το κείμενο τη μερική συμφωνία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη θέση του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση από τα θέματα που άπτονται τη ε, αρμοδιότητα ΛΥΜΠΕ. Έχουμε το πρόγραμμα δικαιοσύνη και το πρόγραμμα δικαιωμάτων και αξιών και είναι σε αυτή την κατάσταση. Ξέρετε ότι σήμερα εγκρίναμε τι μερικέ συμφωνίε. Ε, Επομένω, ε, θα πρέπει να δούμε αν την 1η Δευτέρα Απριλίου θα προχωρήσουμε με την επικύρωση. Θέλω βέβαια να συγχαρώ όλου για την επίτευξη των συμφωνιών αυτών. Τώρα, η απόφαση εξαρτάται και από την ε, επιστολή του Συμβουλίου που επιβεβαιώνει τη μερική συμφωνία. Έχουμε αυτή την επιστολή όπως ακούσαμε πριν. Και θα τα βρείτε όλα αυτά σε αντίτυπα στα έγγραφα στο φάκελό σα. Τώρα, σε ό,τι αφορά άλλα ζητήματα, έχει ολοκληρωθεί στην πρώτη ολομέλη του Μαρτίου η τοποθέτησή μα σε πλαίσιο τη πρώτη ανάγκη. Δεν έχουμε μέχρι στιγμή το Συμβούλιο εντολή για τι διαπραγματεύσει. Οπότε, εκτός αν υπάρχουν τεχνικοί λόγοι ε, προς τούτο, οι θέσεις που εγκρίναμε στην πρώτη ανάγνωση της τρέχουσας θητείας θα είναι η αφετηρία για την επόμενη θητεία. Σε ό,τι αφορά ε, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης, το Ταμείο Στερικής Ασφάλειας και το Ταμείο Διαχείριση Συνόρων και Θεωρήσεων. Η Κομισιόν προτείνει κάποιες διατάξεις στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού που θα επηρεάσουν τα εν λόγω ταμεία. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ε, με το Συμβούλιο και αυτό το γενικό κανονισμό στις σαφές πως η συμπερίληψη των ταμείων της ΓΔ Home στο πλαίσιο της λεγόμενης συμφωνια σχέσης άρθρο 7 είναι ένα σημαντικό σημείο συζήτηση. Θα θέλει λοιπόν το Κοινοβούλιο διατάξει τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση να είναι πιο ενισχυμένε. Όμω το Συμβούλιο θέλει τα ταμεία του Home να εξαιρεθούν αυτή τη διάταξη για λόγου απλούστευση. Προ το παρόν, εξελίσσονται, είναι σε εξέλιξη διαβουλεύση μεταξύ των εισηγητών ε, από τη Ρέγκη, είναι η κυρία Κρέλα από των Σοσιαλιστών και ο κύριος Νοβάκοφ από το ΕΛΚΑ. δεν επικοιτά απόφαση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να εγκρίνει την εντολή για το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Κατά πάσα πιθανότητα οι διαπραγματεύσει θα συνεχιστούν μετά τι εκλογέ. Τώρα, μια ενημέρωση για τι εξέλιξει του Συμβούλου ό,τι αφορά τον κανονισμό για το ΠΔΕΛΤΑΠΗ και τα αριθμητικά στοιχεία. Μα ενημέρωσε η Επιτροπή Προπολογισμών ότι δεν υπάρχει πλέον πίεση χρόνου, γιατί δεν ε, έχει κανένα σχέδιο το Συμβούλιο να εγκρίνει τη θέση του πριν από τι εκλογέ. Μόνο μάλλον τον Οκτώβριο του 2019. Περιμένει βέβαια να έχει εγκρίνει το Συμβούλιο του κανονισμού, βασικού κανονισμού για το πι-δελ-τα-πι στα τέλη του 2019, αλλά μάλλον τη διαδικασία έγκριση θα ολοκληρωθεί το 2020, γιατί θα ήθελε να διαπραγματευτεί το Κοινοβούλιο πριν δώσει τη σύμφωνη γνώμη του, που σημαίνει ότι ε, η Ρουμανική Προεδρία δεν θα δημοσιοποιήσει ε, κάποια επικαιροποιημένη εκδοχή του διαπραγματευτικού κουτιού και εμεί θα ξέρουμε για τα τομεακά προγράμματα, τα χρήματα που θα έχουμε διαθέσιμα το νωρίτερο στα τέλη του φθινοπόρου. Αυτό είναι πολύ δύσκολο όταν έχουμε θέματα για τα οποία το ποσό που διατίθεται θα επηρεάσει ιδιαίτερα τη δομή ενό ταμείου ενό προγράμματο. Όπω παραδείγματο χάρη το πρόγραμμα δικαιωμάτων και αξιών. Σας εξήγησα λοιπόν ε, περί τίνος πρόκειται, σας έκανα αυτές τις ε, τρεις ε, παρουσιάσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια. διά Διάθ Ντεμέρα, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση αυτή κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω μια προειδοποίηση. τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά η Europol και άλλες ε, φορείς ασφαλείας, ε, αναθέσαμε νέες αρμοδιότητες και νέα καθήκοντα. Η εμπιστοσύνη των κρατών ε, στην Europol έχει αυξηθεί σημαντικά και η Europol επεξεργάζεται ένα πολύ μεγαλύτερο, εκθετικά μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων και υπάρχουν όλο και περισσότερα αιτήματα επιχειρησιακής και αναλυτικής στήριξης, όπως γνωρίζετε. Η πρόταση για το πιδέλτα ποιος έχει αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τα κονδύλια για τη Europol, κατά μένα επαρκής. Και θα σημάνει ουσιαστικά μείωση του προβλησμού της Europol για την ε, εν λόγω περίοδο ε, σε σύγκριση ε, με την τρέχουσα και αυτό θα δημιουργήσει δυσκολίες στο να διατηρήσει τις επιδόσεις της Europol αλλά θα παρέχει μειωμένη επιχειρησιακή υποστήριξη στα κράτη-μέλη. Κατ' Δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτήν ε, την δημοσιονομική πρικοδότηση και ως κοινοβούλιο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, ε, ελπίζω ότι μπορούμε ως κοινοβούλιο να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τα κονδύλια τα γενικά κονδύλια, έχουμε αύξηση από 5 σε 7. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική ασφάλεια, από την ασφάλεια και τους πολίτες πάμε στην ασφάλεια και στην άμυνα. Η νέα δομή του πλαισίου δεν προβλέπει μεταφορά προπολογισμού ε, στην στα θέματα τζάι, εσωτερικής ε, πολιτικής, εσωτερικών θεμάτων και δικαιοσύνης. Στο παρελθόν ήταν δυνατόν μέρος του προϋπολογισμού που δεν είχε εκτελεστεί από τη Frontex ε, να ε, μπορεί να εκτελεστεί. Εδώ έχουμε 1,1 δις για τις διάφορες, για τους διάφορους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται με τι ασφάλειε. Για την Ευρωπόλη έχουμε 937 δι που προβλέπονται για την επόμενη περίοδο. Και αυτά δεν επαρκούν για το 2021-2027. Η Κομισιόν θα ε, μειώσει λοιπόν σημαντικά τον προπολογισμό τη Europol. Να σα δώσω και ένα παράδειγμα. Το 2021 προπολογισμό που προβλέπεται είναι 126 εκατομμύρια, ενώ το 19, το τρέχον έτος, ο προπολογισμό είναι 138 εκατομμύρια, που σημαίνει 12 εκατομμύρια λιγότερα. Ε, Επομένω, βλέπετε, αυτό θα έχει δεινέ συνέπειε για την ασφάλεια των Ευρωπαίων, εφόσον παραμείνει έτσι ο προπολογισμό. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Υποστηρίζω τα ζητήματα που αναφέρατε. και τα οποία τέθηκαν και στην πρόσφατη συνάντηση της JPSG. Να πω τώρα στα υπόλοιπα μέλη ότι δεν συζητούμε απλώς περισσότερα χρήματα. Πρόκειται για σημαντικές πιέσεις προς την Ευρωπόλ. Τους έχουν ζητηθεί λοιπόν να αναλάβουν πολύ περισσότερα καθήκοντα. Τα θεσμικά όργανα τους έχουν ζητήσει χωρίς να τους προσφέρουν την αναγκαία χρηματοδότηση. αυτού του είδους η λεπτομερής παρέμβαση που κάνατε έγινε και στην JPSG. Ευχαριστώ λοιπόν. Πρώτα κυρία Σίπελ και θα ακολουθήσει η κυρία Ευχαριστώ αγαπητέ πρόεδρε. Να προσθέσω κάτι στα όσα είπε ο κύριος Τιάθτε Μέρα. Το πρόβλημα είναι, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο μέσα στις ίδιες τις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι χώρες μέλη ζητούν όλο και περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και αυτό έχει καλώς καταρχήν. Το υποστηρίζω και εγώ. Όμως οι χώρες μέλη δεν προσφέρουν και την αναγκαία χρηματοδότηση και όχι μόνο για θέματα εντό των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ αλλά και αλλού όπου προστίθεται διαρκώς καθήκοντα, αποστολές αλλά δεν χρηματοδοτούνται. Και τώρα και για το επικείμενο Brexit, το οποίο δυστυχώς οφείλω να επαναλάβω, θα έχουμε ένα μεγάλο κενό στους επόμενους κοινοτικούς προϋπολογισμούς. Άλλο είναι το τι μπορούμε να κάνουμε εντό του υφιστάμενου προπολογισμού και άλλο είναι να μιλήσουμε για πρόσθετο νοπό χρήμα, διότι αλλιώ θα θα πάντοτε να κρίνουμε πού θα περικόψουμε κάποιες δαπάνες παραβιάζοντας έτσι την υποχρέωσή μας να φροντίζουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και που θα δώσουμε αλλού. Πρέπει να γίνει η συζήτηση για το πώς μπορούμε να περιλάβουμε περισσότερα κονδύλια στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, ώστε να εκτελεστούν όλε οι αποστολέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση που επιθυμούν να δουν οι Ευρωπαίοι πολίτε. Συμφωνώ μαζί σα, λέει ο Πρόεδρο. Βλέπω και τον μεγάλο κατάλογο ονείων της ε, JPSG και του Συμβουλίου, η Ευρωπόλ δεν είναι και κανένα τεράστιο οργανισμό. Δεν καταλαβαίνει τι πραγματικέ διαστάσει ορισμένοι. Ο προπολογισμό πρέπει να ανταποκρίνεται στι προσδοκίε. Και ο ίδιο ο διευθυντή του είναι ανήσυχο. Αντιλαμβάνεται ότι η Ευρωπόλ δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και αυτό ισχύει και για άλλου οργανισμού. Το παράδειγμα αυτό τη Ευρωπόλη είναι καλό. Η κυρία Χολμάιερ. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απολύτω με τον κύριο Ντία Στεμέρα και προσυπογράφω ρητά. Τα όσα είπε είναι απολύτω θεμελιωμένα. Με την Ειδική Επιτροπή του Αγώνα κατά τη Τρομοκρατία αποφασίσαμε ότι θέλουμε να επιταχύνουμε, για παράδειγμα, διαδικασία διαδικασίε ανταλλαγή πληροφοριών η Ευρωπόλ με το παλαιό τη σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλέον στις απαιτήσει που ε, προβάλλει το Κοινοβούλιο και στην ίδια την εντολή. Και στον επόμενο προπολογισμό του 2020 δηλαδή δεν προβλέπονται ούτε καν χρήματα για την ίδρυση του κατάλληλου συστήματος ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων. Άρα, εφόσον μεταφέρονται καθήκοντα σε έναν και μάλιστα σοβαρότατα καθήκοντα τα οποία το ε, και τη ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών, πρέπει αυτά να χρηματοδοτούνται επαρκώ. Και δεν μιλούμε για εκατοντάδε εκατομμύρια. Μιλούμε για ίσω πρόσθετα κονδύλια 10-20 εκατομμυρίων έτος. Δεν μιλούμε δηλαδή τώρα για τάξει μεγεθών που θα διαρρήξουν τα όρια του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Μιλούμε για λογικά και σχετικά μικρά ποσά επισημαίνω ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Eurojust καθώ και στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα, του Ευρωπαίου συγγνώμη, Εισαγγελέα, όπου δεν λειτουργεί καλά η συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών. Ίσως ω Κοινοβούλιο πρέπει να φροντίσουμε ώστε και οι τρει προαναφερθέντες οργανισμοί να έχουν επαρκή, δεν μιλώ για τεράστια ποσά και πάλι, αλλά να είναι επαρκώς χρηματοδοτούμενοι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά του. Πρόεδρος σωστή, πολύ ε, σημαντική παρέμβασή σας για να καταλάβουν οι συνάδελφοι πόσο ε, στενή είναι η επαφή με το προσωπικό της ε, Eurojust. Οι αριθμοί τους είναι μικροί, όμως η προσφερόμενη προστιθέμενη αξία είναι σημαντική από τις δραστηριότητε τους. Η Eurojust είναι ο διαδικαστικός βραχίωνας. Όμως είναι λίγοι για τη δουλειά που τους έχει ανατεθεί. Μικρές αυξήσεις λοιπόν του προπολογισμού τους αποδίδουν μεγάλη αξία. Και η Eurojust λοιπόν είναι ένα καλό παράδειγμα. Πρέπει όμως να διορθώσουμε την κατάσταση και για Ευρωπόλ και για ε, Eurojust και νομίζω ότι με τις παρεμβάσεις σας ε, περιγράψατε την θέση μας. και θα μεταφέρω το περιεχόμενο των παρεμβάσεων σας και στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπόλ. Άλλος κανείς παρακαλώ θέλει να παρέμβει για θέματα προπολογισμού. Γεράρ. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Εγώ υποστηρίζω απολύτως τα όσα λέχθηκαν έως τώρα από τους συναδέλφους μου και τα οποία επαναλάβατε. Πρέπει να προβλεφθούν τα αναγκαία κονδύλια ώστε οι οργανισμοί να μπορούν να εκτελούν σωστά τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από Κοινοβούλιο και από Συμβούλιο. Άρα συμφωνώ απολύτως με, την, με το αίτημα αύξησης των κονδυλίων για να μπορούν να τα αποκρίνονται στα καθήκοντά τους. Ευχαριστώ Ζεράρ, πραγματικά με τον τρόπο αυτό ολοκλήρωσες ε, ε, τον αριθμό των ε, σημαντικών αυτών παρεμβάσεων θα είδατε ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα στέρεο γραφείο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό με τις, ε, και να ανταποκρίνει τι προσδοκίε αυτέ που είναι υψηλέ, εάν δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση. Καλώ λοιπόν. Ας προχωρήσουμε τώρα στη μελέτη. το υπαριθμό 11 δηλαδή, που είναι μελέτη για θέματα παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, τα περίφημα fake news, άλλοι τρόποι επηρεασμού της κοινή γνώμης. Δυστυχώς αναπτύσσονται ιδιαίτερα αυτά τώρα που πλησιάζουμε σε ευρωεκλογέ. Πολλοί έχουν εργαστεί για το θέμα αυτό σε ακροάσεις ε, με εκπροσώπους του Facebook και άλλα σχετικά. Και πρόκειται τώρα για την παρουσίαση μελέτης που ανέθεσε το Τμήμα Πολιτικής. Ε, νομίζω είναι η κυρία Μπάγερ μαζί μας, η οποία θα προχωρήσει σε παρουσίαση. Και πιστεύω θα τη βρείτε ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Είναι τιμή μου που μπορώ να σας παρουσιάσω αυτή την ε, μελέτη που έχει ως ερώτημα πώς η παραπληροφόρηση και η προπαγάνδα επηρεάζει τη λειτουργία του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της εκπονήθηκε από έξι εξαίρετους συντάκτες η έκθεση αυτή και είχαμε και τρεις άλλους που συνεισέφεραν. Την αναθεώρησαν δε δύο ανεξάρτητοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες ως εξωτερικοί αναφερτές αλλά και άλλοι ε, από την υπηρεσία έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα νομίζω ότι είναι μια διεξοδική έρευνα και ένα νέο δε πεδίο ερευνητικό χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι και μέσα. Υπάρχουν και περισσότεροι που ασχολούνται με το θέμα αυτό από τότε που έχει ε, κινήσει και το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες ε, σε ό,τι αφορά ε, το περιεχόμενο. Θα σας πω απλά ποια είναι η δομή και θα εστιάσω στα κυριότερα. Πρώτα απ' όλα, ε, πεδίο εφαρμογή και ορισμός. Τι εννοούμε με τον όρο ε, παραπληροφόρηση το πρώτο. Έπειτα αναφέρονται τα βασικά, ε, τα ορόσημα της έξτρα τη παραπληροφόρηση, τι δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ω πρόβλημα στι δημοκρατικέ κοινωνίε. Έπειτα μιλούμε για κάποιε θεωρητικέ έννοιε και υποθέσει ε, που εξηγούν ε, το μεταλλασσόμενο αυτό περιβάλλον ε, στα μέσα ενημέρωση και στι κοινωνίε και επίση μετά η έκθεση αναλύει το πώ επηρεάζεται η δημοκρατική διαδικασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου στι ευρωπαϊκέ χώρε. Αναλύει επίσης ε, το νομικό πλαίσιο, δηλαδή τους υφιστάμενους νομικούς κανόνες και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μιλούμε επίση για νομικού κανόνε που έχουν συνταχθεί τα δύο-τρία τελευταία χρόνια για την καταπολέμηση του φαινομένου τη παραπληροφόρηση ε, και κρίνουμε την αποτελεσματικότητά του. Επιπρόσθετα γίνεται λόγος ε, για τις μελλοντικέ αποτρεπτικές ε, τεχνολογίες και την έρευνα και τα πορίσματά της. Δημόσια γλώσσα, ε, δημόσιος διάλογος. Είναι ο πυλώνας της δημοκρατίας και βλέπουμε ότι η γλώσσα αλλάζει ε, στην εποχή του διαδικτύου. Πρώτα απ' όλα όλοι ε, περιλαμβάνονται, και αυτοί που μάλλον κανένα δεν, δεν έχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιος θεματοφύλακας, κάποιος ε, κλειδοκράτορα. Ο καθένα μπορεί να έχει πρόσβαση. Δεν χρειάζεται να είναι καν ε, κάποιος ε, ε, Μπορεί και ένας αναλφάβητος ε, να έχει πρόσβαση. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και τεχνητέ μέθοδοι ε, διάδοσης για την προώθηση περιεχομένου. Χρειάζεται απλά κάποιο να έχει οικονομικά μέσα στη θέση του. Το συμπεριφοριστικό μάρκετ τεχνολογία χρησιμοποιούνται επίσης για να ε, στοχευθεί ε, κομμάτι του πληθυσμού και να μεταδοθούν μηνύματα με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο με την λεγόμενη μεροληψία που οδηγεί σε πόλωση του ακροατηρίου καθότι έχουμε διεύρυνση ε, του, της δημόσιας σφαίρας. Και αυτή η νέα δημόσια σφαίρα ε, είναι πιο συμμετοχική από ό,τι πριν, αλλά τα μηνύματα τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα, στοχευμένα μεταδίδονται με ταχύτητα του φωτός, ενώ επιχειρηματολογία, λογικές ε, επιστημονικές πληροφορίες ε, μένουν πίσω. Έχει αυξηθεί δηλαδή η διάσταση μεταξύ κάποιων πιο επιστημονικών επιθεωρήσεων και των λαϊκών μίντια. Ε, στην έρευνά μας διαπιστώσαμε δύο παράγοντες που οδηγούν ή που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των εκστρατιών παραπληροφόρησης πλουραλιστικό υπόβαθρο. Τα μη πλουραλιστικά ε, είναι στόχος ε, πιο εύκολος, γιατί αυτά τα κροατήρια δεν έχουν τη δυνατότητα να διασταυρώσουν πληροφορίες. Και επίσης το επίπεδο διοργάνωση εκστρατείας παραπληροφόρησης σποραδικά συμβάντα έχουμε, δημοσιεύονται από μικρά ε, μέσα. Απ' την άλλη έχουμε όμως ε, ε, συντονισμένες και πολύ καλά χρηματοδοτούμενες εκστρατείες. Εξετάζοντας τώρα τα θεμελιώδη και πώς επηρεάζονται από αυτό το φαινόμενο, εντοπίσαμε τρία βασικά ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία πλήττονται άμεσα από την παραπληροφόρηση. Το πρώτο είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια που οδηγεί και σε άλλα προβλήματα όπως ε, στην έλλειψη ιδιωτικότητας ή ε, ελευθερίας έκφρασης. Έχουμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης που οδηγεί σε παραπληροφόρηση και προσανατολή στην κοινή γνώμη. Ε, θεωρούν ότι πρόκειται για ανθρώπου ενώ δεν είναι έτσι και με την τεχνολογία μπορεί κανείς τα ευάλωτα σημεία του καθενός ε, να τα ε, ευαισθητοποιήσει και να επηρεάσει με βάση τις φοβίες ε, ή τις ανησυχίες του καθενός. Επίσης, το δεύτερο είναι η ιδιωτικότητα και το δικαίωμα προστασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα. Με μικροστόχευση πλήττεται αυτή, αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα. Με ένα περιορισμένο κροατήριο στο οποίο υπάρχει ένα μήνυμα ε, που θεωρεί ο αποστολέας του μηνύματος ότι θα δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το μήνυμα. Οι ε, αλγόριθμοι βοηθάνε πολύ και έχουμε συνεχής προσαρμογής σε προσαρμογές και τελειοποίηση των αλγορίθμων και των σχετικών τεχνολογιών για το σχεδιασμό ε, εξατομικευμένων και πολύ καλά προσαρμοσμένων εκστρατιών, μπορεί να είναι πορικές ή πολιτικές. βασίζεται στα ευάλωτα σημεία και αξιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για να εκμεταλλευτεί ακριβώς αυτά τα ευάλωτα σημεία. Λοιπόν, πέρα από θέματα προστασίας των δεδομένων, αυτή η μικροστόχευση ε, κατακαιρματίζει την κοινή βάση πληροφόρησης για το δημόσιο διάλογο. Και έτσι δεν μπορεί το κοινό να διαμορφώσει μια ενημερωμένη άποψη που να βασίζεται σε στοιχεία αυτή. Η μικροστόχευση λοιπόν έχει διπλή αντική επίδραση. Πρώτα απ' όλα θίγει τα άτομα αυτά στα οποία απευθύνεται, αλλά και αυτοί οι οποίοι δεν λαμβάνουν τα μηνύματα αυτά, δεν γνωρίζουν τι μηνύματα λαμβάνουν οι συμπολίτες τους. Για παράδειγμα έτσι, τα πολιτικά κόμματα στοχεύουν ε, διαφορετικά κοινά και, να, και στέλνουν ακόμη και αντιφατικά μηνύματα στους μεν σε σχέση με τους δε και έτσι να ε, μεγιστοποιήσουν την απήχησή τους. Επίσης, ε, η μικροστόχευση βασίζεται σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Αυτό μας ανησυχεί από πλευράς προστασίας των δεδομένων. Και το άλλο είναι η ε, ελευθερία έκφρασης και η αντική πλευρά η ελευθερία να λαμβάνεις μηνύματα. Η ε, ψεύτικη ενημέρωση δεν είναι παράνομη από, το, από μόνη της, αλλά εάν ένα ε, περιβάλλον ε, κατακλείζεται από παραπληροφόρηση, η βασική αιτία ύπαρξης των μέσων παραβιάζεται. Είναι συστημική παραβίαση της ελευθερίας των μέσων που είναι τμήμα της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας να λαμβάνεις ενημέρωση που είναι βασικό δικαίωμα των πολιτών για να λαμβάνω αποφάσεις με τα λόγου γνώσεως. Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα αλληλοσυνδέονται εν γενός και αλληλοεξαρτώνται. Εάν θυγεί το ένα, θύγεται συνολικά το σύστημα. Το τρίγωνο αυτό. Μιλήσαμε για την ελευθερία έκφραση και την ελευθερία να ενημερώνεσαι. Εάν θυγεί αυτό, τότε η ενημερωμένη συμμετοχή στις εκλογές επηρεάζεται και αυτός είναι πυλώνας της δημοκρατικής δυνατότητας λήψης αποφάσεων. Αν σε ένα κράτος μέλος θυγούν αυτά, θίγεται παντού στην Ένωση. Γιατί οι πολίτε τη Ένωση είναι πολίτε, συγγνώμη, πολίτε του κράτου μέλου αυτού είναι και πολίτε τη Ένωση. Και ο μηχανισμό λήψη αποφάσεων τη Ένωση σε κάθε κράτο μέλο θίγεται. Αν έχουμε δημοκρατικέ εκλογέ, για παράδειγμα ευρωεκλογέ σε ένα κράτο μέλο, εάν επηρεαστούν από αυτή την ε, προσπάθεια επηρεασμού τη προεκλογική εκστρατεία, αυτό ε, μπορεί να θίξει την νομιμοποίηση συνολικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ έχουμε ένα πίνακα. Πώς λοιπόν ο επηρεασμό των δημοκρατικών διαδικασιών και η στρέβλωσή τους και η ακύρωση της δημοκρατίας ε, αλλοσυνδέονται. Και τι μπορεί να κάνει η Ένωση γι' αυτό. Εδώ στα αριστερά η στήλη δείχνει πώς επηρεάζονται όλα αυτά και αν γίνονται σεβαστά ή αν γίνεται προσπάθεια στρέβλωσής τους και οι γραμμές δείχνουν αν διατηρείται ή αν ανατρέπεται η δημοκρατία και έχουμε διάφορα ε, υποθετικά σενάρια το πρώτο είναι το α ας πούμε όταν όλα είναι τέλεια το β είναι όταν οι μέθοδοι της ε, δημοκρατίας φύγεται και ε, κερδίζουν αυταρχικές ε, δυνάμεις εκλογές. Ναι, μεν τυπικά γίνεται σεβαστή δημοκρατική διαδικασία, αλλά προκύπτει αυταρχική κυβέρνηση, η οποία μετά μπορεί να ανατρέψει τη δημοκρατία. Άρα πρέπει να ισχύσουν οι εποπτικές αρχές της Ένωσης. Και στο σενάριο C, η δημοκρατική διαδικασία στρεβλώνεται. Για παράδειγμα, με αλλαγή των εκλογικών περιφερειών, με παράνομη χρηματοδότηση της προηγής εκστρατεία. Το αποτέλεσμα δεν ε, ακυρώνει τη δημοκρατία και σε αυτή την περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει αν τα διαδικαστικά θέματα είναι αρκετά σοβαρά, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ελέγχου εάν ε, το άρθρο 2 ε, έχει γίνει σεβαστό. Και το σενάριο Δέλτα. Σαφής περίπτωση ενεργοποίησης του μηχανισμού του άρθρου 2 όταν και η διαδικασία έχει στρεβλωθεί και το αποτέλεσμα των εκλογών μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της δημοκρατίας. Οι συστάσεις μας περιέχονται σε δύο δέσμες. Πρώτον, να ενισχυθεί η δημοκρατική αντοχή και ένα δεύτερο. Για το πρώτο λοιπόν, η μελέτη μας εξετάζει τι εννοούμε με τον όρο αντοχή της δημοκρατίας. Χρησιμοποιούμε και τον όρο ενεργή δημοκρατία. Και ε, ε, εξηγούμε και ποιες είναι οι βασικές αρχές αυτής της ιστορικής ε, ε, έννοιας. Εξηγούμε τι σημαίνει αντοχή, ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, και ποια μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τα μέσα αυτά είναι προληπτικά. Μπορούν να ε, προλάβουν την ε, διάβρωση και ανατροπή της δημοκρατίας και ακύρωση της δημοκρατίας και ε, εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, εάν ακυρωθεί η δημοκρατία είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει. Εδώ λέμε πώς θα ενισχύσουμε τη δημοκρατική αντοχή. Τέσσερα σημεία για τα οποία έχουμε κάνει συστάσεις και εν ώψη των ε, επερχομένων ευρωεκλογών. Και πιο μακροπρόθεσμα. Προτείνουμε να υπάρχουν αυστηρότεροι κανόνες, οι οποίοι να είναι ουδέτερα σοφρά τις πλατφόρμες για την ε, πολιτική διαφήμιση, που να είναι αναρμονισμένα μεταξύ κρατών μελών. Από αυτό χρειάζεται και ουσιώδης μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατιών για να υπάρχουν σαφέστεροι κανόνες, πιο διαφανείς κανόνες. Γιατί αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, μια χρόνια ασθένεια της δημοκρατίας μας. Το τρίτον είναι να προστατεύουμε με αυστηρότητα τα προσωπικά δεδομένα. Ο γενικός κανονισμός ε, είναι βασικό εργαλείο, αλλά δεν ε, έχει ολοκληρωθεί η εργασία. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο κανονισμός για την ή ε, προστασία των, της ιδιωτικής σφαίρας και οι κανόνες αυτοί να εφαρμόζονται και να συμπληρωθούν με πρακτικές φιλικές προς το χρήστη. Γιατί η εφαρμογή του γενικού κανόνα οδηγεί σε μια κόποση με την ανάγκη να δίνει συνέχεια τη συνένεσή σου και κυρίως στις ε, περιφερειακές περιοχές και γεωγραφικά και κοινωνικά πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Να ενημερωθεί το κοινό, για τις αξίες της Ένωσης, για τη δημοκρατία, για το πώς πρέπει να διοργανώνονται οι εκλογές, να ευαισθητοποιηθούν για την παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα. Και η ποιότητα αυτών των ε, προγραμμάτων πρέπει να ελέγχεται από την Ένωση και τα μέσα και τους ε, θεσμούς της Ένωσης. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά σε τοπικούς φορείς. Τα προγράμματα ενημέρωση για τα θέματα αυτά θα πρέπει να συμπληρωθούν με εκπαίδευση των διδασκόντων Επίσης, ε, να προσπαθήσουμε να φτάσουμε και σε κοινότητες ε, όπου δεν έχουμε φτάσει ακόμη. Επίσης, να υπάρχουν αρχές για ε, δεοντολογική χρήση των κοινωνικών μέσων, όχι μόνο για την παραγωγή περιεχομένου, αλλά και για το πώς γίνεται το like και τα λοιπά και πώς θα μοιραζόμαστε με άλλους. Πρέπει να δημιουργήσουμε επανέλθουμε, να επανέλθουμε πρέπει να δημιουργήσουμε πυλώνες εμπιστοσύνης. Πυλώνες λοιπόν εμπιστοσύνης προς τα μέσα, το περιβάλλον των μέσων και κυρίως τα δημόσια μέσα. Να δούμε αν τα δημόσια μέσα πρέπει να ε, εξυπηρετούν πραγματικά τις ανάγκες του κοινού. Δεν είναι δυνατόν δημόσια μέσα να είναι φορείς παραπληροφόρηση. Πρέπει να τα ελέγχει η Κομισιόν αυτά. Και αν διαπιστώνει ότι κρατικά μέσα δεν βοηθούν την ενημέρωση του κοινού, αλλά είναι όμοιροι των κυβερνήσεων ή πολιτικών κομμάτων, τότε δεν θα πρέπει να εγκρίνεται η εξαίρεση όσον αφορά τη χορήγηση κρατικών βοηθειών. Επίσης πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες για τη συγκέντρωση ιδιοκτησία μέσων. Και αυτό πρέπει να εφαρμοστεί και για τις πλατφόρμες και άλλες εταιρείε ιδιοκτησίας μέσων. Πολλοί έλεγχοι πρέπει να γίνονται για να διατηρήσουμε την πολυφωνία των μέσων. <clears throat> Θα πρέπει να είναι τμήμα αυτό του μηχανισμού επιτήρησης για το κράτος δικαίου, για να αποφύγουμε πισωγυρίσματα. Όσον αφορά τις πλατφόρμες, έχουμε μια σειρά από το κύριο είναι όχι να προσπαθούμε να κάνουμε λογοκρισία των ψευδών ειδήσεων, αυτό δεν λειτουργεί. Αλλά να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο για να ακούγονται όλες οι φωνές. Δεν θέλουμε να ε, απαγορεύει το κράτος ε, τις ε, ψευδείς ειδήσει, αλλά να επηρεάζει θετικά τη διάδοση των σωστών πληροφοριών. Για παράδειγμα, το επιχειρηματικό μοντέλο είναι πώς ε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε για χρηματικό όφελο στα προσωπικά δομένα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Τώρα, συστάσει για τις πλατφόρμες. Κυρίως το 2 σε αυτό τον κατάλογο. Θα πρέπει να απαιτείται οι κυρίαρχες πλατφόρμες να έχουν μια ουδετερότητα στις υπηρεσίες και να μην κάνουν διακρίσεις και όσον αφορά το περιεχόμενο και τους χρήστες με βάση τις ε, πολιτικές τους ή άλλα προστατευόμενα χαρακτηριστικά. Για να συνοψίσω. Η μελέτη μας περιέχει πολλές συστάσεις. Σας ε, συστήνουμε να τις διαβάσετε, αλλά να σταθώ σε μερικά σημεία που είναι τα βασικότερα. Μακροπρόθεσμα που θα αλλάξουν πραγματικά την κατάσταση ριζικά, να αλλάξει γενικά το πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα να αυξηθεί, να δημιουργηθεί καλύτερα η αντοχή της δημοκρατίας για να μετωπιστεί η παγκόσμια τάση των λαϊκιστικών ε, αυταρχικών τάσεων. Και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις μελλοντικέ τεχνολογίες. Οι τεχνολογίες θα βασιστούν όλο και περισσότερο στην ε, εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και θα οδηγήσουν σε ουτοπικές κοινωνίες. Και πρέπει να αναθεωρηθεί και ο τρόπος ε, διεξαγωγής των πολιτικών εκστρατιών. Αυτό είναι μακρόπνο έργο. Η Ένωση είναι σε θέση να δράσει για τα θέματα αυτά πολύ καλύτερα από τα κράτη-μέλη. Πρώτα απ' όλα η χρηματοδότηση των εκστρατιών πρέπει να ρυθμίζεται. Δεύτερον, να είναι δεοντολογικές αυτές οι εκστρατείες, να είναι δίκαιες, να είναι αυτορυθμιζόμενες οι πρακτικές αυτές από όλους. Αυτό θα το εκτιμούσαν και οι ψηφοφόροι. Γι' αυτό χρειάζονται προγράμματα ε, κοινωνικής ενημέρωσης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Υπάρχουν και άλλες, ε, και άλλα αντίγραφα όπως αυτό που ε, σας έδειξα κρατώντας τα χέρια μου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάγερ, ευχαριστώ και τα μέλη που παρακολούθησαν την ε, ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ελπίζω ότι είναι χρήσιμη για τους συναδέλφους. Παρακαλώ ερωτήσεις. Μπάρμπαρα Σπινέλη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση καθώς και για την μελέτη. Βέβαια δεν μπόρεσα να τη διαβάσω όλη. Ε, τη διάβασα διαγωνίως, όπως ε, λένε. Όμως, συμφωνώ με πολλές από τις συστάσεις που έχετε περιλάβει σε αυτήν και τονίζω ιδίως κάποια γεγονότα που γνωρίζω. Όταν ήμουν εισηγήτρια, για την ελευθερία του τύπου και τότε ε, στην εργασία μου είχα επιμείνει σε ένα θέμα ότι υπάρχει κινδυνολογία για την παραπληροφόρηση στην επιγραμμικά στο διαδίκτυο δηλαδή και εν μέρει αυτό είναι θεμητό Και το θέμα της παραπληροφόρησης θίγει ακόμα και μεγάλες έγκυρες εφημερίδες. Ήδη από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και από τον πόλεμο της Κορέας πιο συγκεκριμένα. Και είναι πολύ έντονο. Έχω υπάρξει δημοσιογράφος και έχω μάθει πολλά πράγματα στη δραστηριότητα αυτή. Το leitmotiv του Economist ήταν να υπεραπλοποιούν και να υπερβάλλουν. Όταν μιλούν για υπερβολική παρουσίαση πληροφοριών, και στον επιγραμμικό, στην επιγραμμική δημοσιογραφία δηλαδή, ας μην δυσμονούμε ότι αυτό υπήρχε ήδη και το προήγε το ίδιο το περιοδικό Economist. Με ενδιαφέρει το κεφάλαιό σας υπαριθμών 4 για μέτρα που λαμβάνονται σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία για την ε, διαγραφή περιεχομένου από το διαδίκτυο. Εμένα τα μέτρα αυτά μου φαίνονται δυσανάλογα. Αυτά που λαμβάνονται στις ε, χώρες αυτές και είναι λάθος. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από κρατικές αρχές. Ενώ εγώ είμαι υπέρ της αυτορύθμισης. Με αρισχύει πολύ αυτή η task force της ε, Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Δεν πρέπει να υπερβάλλουμε με τα μέτρα αυτά. Τα οποία μου φαίνονται υπερβολικά. Διότι υπάρχει ένα κίνδυνο που έρχεται από πηγέ εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν όμω αναλύσουμε τα αποτελέσματα των ε, ψηφοφοριών, για παράδειγμα, για το Brexit ή τι Αμερικανικέ ή τι Γαλλικέ ή τι Ιταλικέ εκλογέ, λέγοντα ότι τα αποτελέσματα προέρχονται από ρωσικού χειρισμούς δεν υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι τότε που να δικαιολογούν γιατί μια πλειοψηφία Βρετανών ψήφισε υπέρ του Brexit ή γιατί μια πλειοψηφία Αμερικανών ψήφισε υπέρ του Donald Trump. και άλλες ε, δράσεις επιγραμμικά, ιδίως δυσφημιστικές, αποποινικοποιούνται. in your you, Barbara, you did try to cover many of Ξέρω ότι καλύψατε πολλά από τα θέματα αυτά στην έκθεσή σας. Είναι όμως ε, δύσκολο ο τομέας αυτός. Σε ό,τι αφορά τώρα την μελέτη σας, αναφερθήκατε σε ορισμένα από τα κεφαλαία. μεγάλο μέρος από, την, ε, από τις μεγάλες εφημερίδες, από τις ε, ε, μεγάλες οίκους τύπου, δημοσιεύουν τώρα πλέον στο διαδίκτυο, όπως ο οίκος Μέρδοκ. Και από εκεί προέρχονται, όπως Μέρδοκ, Associated Press κλπ. Αυτού του είδους η προσέγγιση αναφέρεται και στην συγκέντρωση του τύπου σε χέρια λίγων ιδιοκτητών, Ωστόσο και ο έντυπος τύπος ακόμη διαβάζεται από πολλούς. Μιλούμε συχνά μονάχα για το προϊόν online και ξεχνούμε την επιρροή στην πολιτική των μεγάλων μαζών που διαβάζουν τον έντυπο τύπο. Δεν ξεχνούμε αυτά ενώ μιλούμε μόνο για Facebook και άλλα επιγραμμικά προϊόντα. Με ενδιέφερε ποια είναι η προσέγγιση σας ως πανεπιστημιακού για αυτή την ικανότητα επηρεασμού. Χθε, για παράδειγμα, προβαίνει σε δήλωση η ε, και η δήλωσή της εμφανίζεται σε προϊόντα μαζικής, μαζικού αναγνωστικού κοινού. Δεν μιλούμε όμως μόνο για προϊόντα online τελικά υπάρχει επηρεασμό τη κοινή νόμη και από τον συνήθι τύπο. Και μιλώ και για online products όπως Daily Mail κλπ. που έχουν τεράστιες δυνατότητες επιρροής. Η κυρία Σαρτζεντίνη Τζούντις. Ευχαριστώ. Κάπως θεωρητικά ήταν αυτά. Μήπως μπορείτε να μας τα πείτε λίγο πιο ξεκάθαρα και να μας δώσετε και παραδείγματα για το πώς καταλήξατε στα συμπεράσματα αυτά. Βλέπω ότι βρέχετε από τη Βουδαπέστη. Ίσως μπορείτε να μας δώσετε ουγγρικά παραδείγματα και μιλούμε και για micro-targeting. Εδώ μιλείτε σε πολιτικού, Δύο μήνε, μόλις μήνες πριν από τι ευρωεκλογέ. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα πράγματα για το πού βάζετε τα όρια. Τα κοινωνικά μέσα είναι εδώ και θα παραμείνουν και διοχετεύουν διαφορετικά μηνύματα σε διαφορετικές ομάδες προσώπων. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που υπερβαίνει τα όρια. Ευχαριστώ, Τζούντιθ. Μπίργκιτ. Σας ευχαριστώ. Ας αρχίσουμε με μια γενική παρατήρηση. Όταν μιλήσατε για καλύτερη νομοθετική ρύθμιση, προστασία δεδομένων και προσωπικής σφαίρας σε ένα κόσμο όπου λίγο πολύ όλα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή. Εγώ τονίζω ότι όντως έχουμε πρόβλημα διότι στην τρέχουσα κατάσταση όταν μιλούμε για GDPR ή privacy και άλλη σχετική νομοθεσία ακούμε ξανά και ξανά και ορισμένες φορές από πολιτικούς αλλά και πολύ συχνά από, τον, ε, από τους άλλους κράτους ότι εμείς από την βιομηχανία κλπ ότι υπερβολικά ρυθμίζουμε, ρυθμίζουμε υπερβολικά για ελεύθερε εκλογέ και για τα οποία μιλήσατε εγώ δεν θεωρώ ότι ρυθμίζουμε υπερβολικά αντίθετα υστερεί χρονικά η νομοθετική ρύθμιση. Το ίδιο για την ελευθερία των μέσων. Τα μέσα, όπως και οποιοδήποτε άλλος χώρος στην ε, κοινωνία μας, δεν είναι από μόνα τους καλά ή κακά. Εξαρτάται πάντως, πάντοτε από το διάφορους παράγοντες. Και τίνουμε να μιλούμε για δημοσιογράφους ε, με καλό εξοπλισμό, μορφωμένους, αλλά βρισκόμαστε και όλο και περισσότερο ε, απέναντι σε μια κατάσταση όπου καθένα μπορεί να βγει και να πει ότι είναι δημοσιογράφος χωρί να διαθέτει τα αναγκαία προσόντα. Και νομίζω ότι και στα μέσα πρέπει να φροντίσουμε ότι οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί γνωρίζουν τους κανόνες, σέβονται τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Και μία από τις διαφορές που έχουμε είναι ότι στον παλαιό ας πούμε κόσμο όπου η έντυπη εφημερίδα όταν έδινε εσφαλμένες πληροφορίες, το κοινό που τα έβλεπε αυτά και αντιδρούσε ήταν σχετικά περιορισμένο. Τώρα στον ψηφιακό κόσμο είτε αρχίσουμε με την παλιά σκοπής εφημερίδα η οποία βεβαίως δημοσιεύεται τώρα και διαδικτυακά οι αντιδράσεις είναι πολύ διαφορετικές. Τώρα για το micro target η μικροστόχευση. Ξαναλέω και πάλι, ότι το πρόβλημα δεν είναι να πούμε ότι η μικροστόχευση από μόνη της είναι καλή ή κακή υπόθεση. Νομίζω ότι τα πολιτικά κόμματα πάντοτε ασκούσαν αυτή την προσπάθεια μικροστόχευσης για να ε, προσεγγίσουν συγκεκριμένες ομάδες δηλαδή. Το πρόβλημα είναι και πάλι ποιος ελέγχει, ποιος ελέγχει αυτούς που προσεγγίζουν το κοινό και πώς αντιμετωπίζει διάφορες μορφές προσέγγισης. Και ευχαριστώ για τις εξηγήσεις και ορισμούς σχετικά με την παραπληροφόρηση, διάφορε μορφέ τη, κακή πληροφόρηση κλπ. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για ποια πράγματα μιλούμε και να βρούμε έναν τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε. Πάντω, η δική μου ερώτηση έχει ω εξή. Στον ψηφιοποιημένο κόσμο που ζούμε, και εμεί οι ίδιε καμιά φορά σκεπτόμαστε με ξεπερασμένου κάπω τρόπου. Ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο, πρώτα, για να εντοπίσουμε την παραπληροφόρηση. Ποιε μπορούν να είναι οι αντιδράσεις πέρα από το πρόβλημα της μικροστόχευσης για να προωθήσουμε ένα αντίθετο μήνυμα. Και τέλος για ενίσχυση της δημοκρατίας και την ενίσχυση της συζήτησης ώστε να γίνουν πιο ουσιαστικές, να ξεφύγουν δηλαδή από τις επικεφαλίδες, διότι οι περισσότεροι ρίχνουν μια ματιά στις, στους τίτλους, διαβάζουν και κανένα tweet και νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα τι πρέπει να κάνουμε στον ψηφιακό κόσμο για να ενισχύσουμε τη δημοκρατία. Που σημαίνει νομίζω ότι χρειαζόμαστε πραγματικές ουσιαστικές συζητήσεις με πραγματικά πρόσωπα σε ένα ε, πραγματικό ε, απτό περιβάλλον. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να μπορούν να αντιδρούν δηλαδή στα διάφορα επιχειρήματα που προβάλλονται από εδώ και από εκεί. Και αυτό επαφίεται νομίζω και στις ε, Δημόσιε αρχέ και στα πολιτικά κόμματα και σε οποιονδήποτε άλλο που πρέπει να προβάλλει ιδέε για να ενισχυθεί η δημοκρατία, να ενισχυθεί η κατανόηση των αρχών τη δημοκρατία και του διαλόγου. Αν ίσω μπορείτε να συμβάλλετε με κάποιε ιδέε ή με κάποιε βέλτιστες πρακτικέ, δεν ξέρω αν στη μελέτη σα έχει περιλάβει βέλτιστες πρακτικέ, γιατί δεν μπορούσα να διαβάσω όλοι. Αν έχετε κάτι τέτοιο όμω θα είναι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο. Ευχαριστώ, Μπίργκιτ. Είναι σημαντική μελέτη για το σημαντικό θέμα. Βλέπετε ότι δρούν οι ευρωβουλευτέ. Αν μπορείτε να απαντήσετε και ιδίω στι πιο συγκεκριμένε ερωτήσει τη κυρία Αργεντίνη. Ευχαριστώ. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις και χαίρομαι ιδιαίτερως που μου τις υποβάλλετε γιατί βλέπω ότι πηγαίνουμε στη σωστή κατεύθυνση με το έγγραφό και με τις συστάσεις μας. Σε ό,τι αφορά την κινδυνολογία και το καινοφανή χαρακτήρα του φαινομένου, νομίζω ότι δεν απλουστεύουμε τα θέμα αυτό που είναι πολύπλοκο σίγουρα. Η παραπληροφόρηση, η κακή πληροφόρηση, είναι κάτι που υπάρχει ε, ίσως από την αρχαιότητα. Από την εποχή του Θεμιστοκλή είχαμε προπαγάνδα και παραπληροφόρηση για να μην μιλήσω τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και επομένως είναι κάτι που προϋπήρχε. Όμως τα δύο-τρία τελευταία χρόνια έφτασε πλέον σε διαφορετικά επίπεδα και είχε και πραγματικό αντίκτυπο στις κοινωνίες. Βέβαια, η σχεση αιτίο-αιτία δεν μπορεί να αποδειχθεί με επιστημονικό τρόπο. Δεν μπορούμε εργαστηριακά να κάνουμε δοκιμές. Παραδείγματος χάρη Αμερικανές εκλογές του 2016 επηρεάστηκαν πραγματικά. Επειδή υπήρξε ρωσική παρέμβαση, αλλά πώς να το αποδείξει κανείς αυτό. Δεν υπάρχει τρόπος και από την άλλη πλευρά αυτό το όλο φαινόμενο ίσως να είναι ε, και διαγενειακό, άρα όχι εφήμερο. Οι ηλικιωμένοι, για παράδειγμα, ανταλλάσσουν 7 ψευδεί πληροφορίε πληροφορίες από τη ΝΕΗ ΕΕ, που σημαίνει ότι οι νέοι είναι πιο καλά εξοπλισμένοι για να αντιμετωπίσουν ε, την ε, παραπληροφόρηση. Είναι η ψηφιακή γενιά. Και ήδη το θέμα αυτό το αντιλαμβάνεται η κοινωνία, οπότε ίσως να υποβαθμιστεί η σημασία του στο μέλλον. Θα δούμε. Η προσπάθειά μας είναι να προσεγγίσουμε τα δομικά ζητήματα του νεομηντιακού περιβάλλοντος και τις δομικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο της δημοκρατίας και των δημοκρατιών. Πώς θα αντιμετωπίσουν οι δημοκρατίες ε, τις προκλήσεις. Το ζήτημα του Brexit, για παράδειγμα, στο έγγραφό μας μιλάμε και για την απογοήτευση των μαζών που πλέον συμμετέχουν ενεργά στο δημόσιο βίο και στο δημόσιο διάλογο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πραγματικά απογοητευμένοι και αν η πολιτική ελίτ δεν καταφέρει να αντιμετωπίσει την απογοήτευση του κόσμου που έχουν πλέον τη δύναμη μέσω των μίντια και μπορούν να επηρεάσουν τη δημόσια γλώσσα, δεν θα αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Τα κοινωνικά μέσα πραγματικά άσκησαν βαθιά επιρροή στη δομή της δημόσιας σφαίρας. Χάμπερμας, ε, και τι λέει ο Χάμπερμας ε, για τη δημόσια σφαίρα. Αλλάζει εντελώς η δομή της δημόσιας σφαίρας. Όλα πλέον είναι πιο διαφανή. Και οι πολιτικές διεργασίες είναι πολύ πιο διαφανείς πλέον. Ε, φαίνεται να είναι πιο κοντά στους πολίτες που όμως δεν μπορούν να τους επηρεάσουν παρόλα αυτά οι απλοί πολίτες και οι απλοί άνθρωποι φαίνεται να έχουν πάρει δύναμη, να ενδυναμώνονται λόγω της συμμετοχής τους στα κοινά δρόμια αλλά δεν φαίνεται να μπορούν να επιτυγχάνουν αλλαγέ. Και υπάρχουν κάποιοι πολιτικοί που υπόσχονται γρήγορε αλλαγέ και να επιτύχουν με τα μηνύματα αυτά που περνάνε. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, το γερμανικό και τον ιταλικό κανονισμό, ε, δεν είναι αποτελεσματική. Συμφωνούμε Ιδίω ο γερμανικό που απευθύνεται συγκεκριμένα ε, σε ρητορική μίσο, σε εγκληματική. Ε, σαν δικαστήρια ε, που αντιμετώπισαν τα εγκλήματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Αλλά είναι εγκληματική ενέργεια ε, και μπορεί να ποινικοποιηθεί η παραπληροφόρηση που δίνεται βάρος εκεί στο γερμανικό κανονισμό. Πρέπει λοιπόν να, ε, να πω ότι αφού μελετήσαμε τα σχετικά κατέληξαμε στο συμπέρασμα ότι μόνο οι διαδικασίες, όχι το περιεχόμενο, γιατί έχουμε τη διαδικασία της, ε, μάλλον έχουμε το πλαίσιο της ελευθερίας έκφρασης. Άρα σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε ορισμένη ε, ρητορική βάση του περιεχομένου της, αλλά του τρόπου διάσωσης. Και εδώ πηγαίνουμε σε κάποιες επιθετικές μεθόδους διάδοσης ε, και μικροστόχευση. Και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Στην εμπορική διαφήμιση είναι μια χρήσιμη τεχνική μικροστόχευση, διότι δεν ε, προσέχουν το άσχετο ή το ακροτήριο στόχος επικεντρώνει την προσοχή τους στο σημαντικό. Και υπάρχει ο εξή απλό κανόνα. Έχουμε το άρθρο 22 του κανόνα για την προστασία των δεδομένων. Κοινή ερμηνεία σε ό,τι αφορά τη μικροστόχευση πολιτικών διαφημίσεων βάσει ευαίσθητων πληροφοριών. Αυτό πρέπει να το δούμε δυνάμει το άρθρο 22. Εκεί εμπίπτει αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επηρεάζεται δηλαδή ε, η απόφαση που λαμβάνουν και από τις διάφορες συνθήκες ε, που ισχύουν για τον εκάστοτε άνθρωπο. Και υπάρχουν συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλίδες, ώστε οι πολίτες, οι χρήστες να μπορούν να διαθέτουν ως θέλουν τα δικά τους προσωπικά δεδομένα και να δίνουν τη συγκατάθεσή τους ενεργά, το λεγόμενο opt-in. Άρα και δεν υπάρχει αντίρρηση, ένσταση. Δεν πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε όμως ως αντικείμενα ε, και να τους ε, στοχεύουμε με αυτές τις μικροστοχευμένες πολιτικές διαφημίσεις, χωρίς να το ξέρουν. Και υπάρχει και το θέμα της διαφάνειας. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση σε μια βιβλιοθήκη διαφημίσεων, σε ένα είδος θετηρίου, πρέπει να ξέρουν τι κριτήρια, ποιος το πλήρωσε, ε, ποιο, ε, που αποσκοπεί, σε ποιους αποσκοπεί αυτή η μικροστοχευμένη διαφήμιση κτλ. Θα πρέπει να έχει επιλογές ο κόσμος που μπορεί να είναι η προσωπική ενημέρωσή του και οι διαφημιστές αυτό μπορούν να το εκμεταλλευτούν για μικροστόχευση. Αλλά πρέπει επίσης να είναι γνωστό που δεν θέλουν. Παραδείγματος ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Είναι κάτι που κανείς μπορεί να το συναγάγει μέσω από τη δραστηριότητα, ε, το περιεχόμενο που βλέπει κανείς ε, ε, και αυτό μπορεί να το ελέγχουν ίσως οι πλατφόρμες και οι πάροχοι, αλλά δεν θα πρέπει να παίρνουν μηνύματα ε, με βάση προσωπικές πληροφορίες τέτοιου είδους συγκεκριμένοι ε, άνθρωποι. Τώρα, το κεφάλαιο μάλλον έχουμε κεφάλαιο συγκεκριμένο για παραδείγματα σε τμήματα και αναχώρα. Για τη δική μου τώρα τη χώρα, την Ουγγαρία, με βάση την επιστημονική έρευνα από το Ίδρυμα τη Οξφόρδης, πρέπει να σας πω ότι είμαστε η μόνη χώρα που η κυβέρνηση βρωμολόγησε ε, την πολιτική κατά της παραπληροφόρησης ε, λόγω του μηδιακού περιβάλλοντος. Σε ό,τι αφορά Scholar το θέμα της αυτορύθμισης. Κατά πόσο υπάρχει λόγος και είναι σκόπιμη αυτορύθμιση. Υπάρχει, ε, υπάρχει θεμητή, υπάρχουν θεμητά επιχειρήματα για την ε, ρύθμιση του μηντιακού περιβάλλοντος, όχι της ελευθερίας έκφρασης βέβαια. Γι' αυτό και είπα ότι προτείνουμε την αρχιτεκτονική του μηντιακού περιβάλλοντος να αυτή να προσαρμοστεί και να επηρεαστεί από τον νομοθέτη και να μην αφαιθεί εξ ολοκλήρου στι ε, διεργασίε τη αγορά που θα καθορίζουν ε, τη δομή τη αρχιτεκτονική και την, ε, το χειρισμό, την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα, δικηγόροι και γιατροί έχουν πρόσβαση και αυτοί σε έναν μεγάλο όγκο πολύ ευαίσθητων και λεπτών πληροφοριών και πρέπει να τηρήσουν το απόρριτο, να είναι χέμηθοι. Γιατί? λόγω της φύσης των υπηρεσιών που παρέχουν. Άρα δεν μπορώ να αποκομίσουν και οικονομικό όφελος από την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Πρόεδρο, στη δική σα ερώτηση, αφήστε τη, ξεχάστε τη, λέει ο πρόεδρο, στη δική μου ερώτηση. Ήταν μια κραυγή απόγνωση κατά έναν τρόπο. Αυτό το Daily Mail που είπα για ότι η Daily Mail δημοσιοποίησε αυτά που πει Mail, αυτό ήταν η κραυγή απόγνωση η δική μου. Τέλο πάντων τα τελευταία 25 χρόνια συμβαίνουν. Δηλαδή η δυσφήμιση των, ε, και η αμάυρωση της Ευρώπης από αυτά τα σφυλάδες, τέλος πάντων. Ευτυχώ έχουν τον Guardian. Και ο Economist, Μπάρμπαρα, καλός είναι και αυτός. Και κατάλαβα αυτό που είπες, ότι ακόμη και ο Economist ε, τα έλεγε αυτά. Πολύ καλό. Εξαίρετη μελέτη, όπως πάντα, Ευχαριστώ να μπορέσουν να το διαβάσουν το έγγραφο. Έχουμε το facebook ε, και όλα αυτά είναι πραγματικά πράγματα που θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον. Ευχαριστώ και ευχαριστώ όλους τους συντάκτες ε, της έκθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Και επαναλαμβάνω, ελπίζω για αυτό το πάρα πολύ κρίσιμο θέμα να αξιοποιηθεί αυτή, το, τα πορίσματα αυτής της έρευνας και της μελέτης σας. Και τώρα θα καλέσω τον Μάικλο Φλάχαρτη ε, να έρθει εδώ. Θα μας μιλήσει ο Διευθυντής της ε, Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Παρακαλώ, ε, μην φύγετε, θα το εκτιμούσα πολύ. Sorry, um, Λοιπόν, Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες αποφάσεις του... της ε, του των Προέδρων, οι οποίες είναι δυσνόητες ο συνήθως, αλλά εν πάση περιπτώσει, προσπαθώ να τις καταλάβω εδώ. Μάικο, πρώτα απ' όλα, Λοιπόν, επειδή είναι τελευταία μας συνεδρίαση, ε, χαίρομαι που συμμετείχα στις εργασίες σας. Έχω επισκεφθεί δύο φορές την υπηρεσία σας και θέλω να το πω τώρα γιατί προς το τέλος δεν υπάρχουν πολλοί θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα όσα έκανες ε, έχει βελτιωθεί πολύ η εικόνα του οργανισμού σας έκανες ό,τι μπορούσες για να έχετε περισσότερες πιστώσεις όλα αυτά είναι αξιοσημείωτα και νομίζω σε ευχαριστώ για αυτά που μας είπες. Και ήταν ε, πολύ δύσκολη περίοδος. Και ευχαριστώ και το προσωπικό σου. Θα το τα πω. Θα μας ενημερώσεις λοιπόν τώρα. Ορισμένοι συνάδελφοι ήρθαν στην υπηρεσία σου στις 25-26 Σεπτεμβρίου ήταν ε, βάση για την παρουσία σου σήμερα εδώ είχατε ένα φόρουμ εγώ συμμετείχα αλλά ως προσθήκη στην αντιπροσωπεία η επίσημη αντιπροσωπεία ήταν η Σεσίλ και κάποιοι άλλοι ήταν πολύ εντυπωσιακή εκδήλωση πραγματικά ασχολήθηκε με την ουσία των καθηκόντων σας. Παρακαλώ κάντε την παρουσίασή σας. Και μετά θα μιλήσουμε και για το φόρουμ. Α, όχι, πρώτα θα πάρει το λόγο η κυρία Κέγκε. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα... Πρώτα απ' όλα θα μας μιλήσει η κυρία Κιέγκε, που ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας, η Σεσίλ Κιέγκε. θα μας παρουσιάσει την επίσκεψη αυτή, την αποστολή και μετά θα μας μιλήσει ο Διευθυντής. Ήταν πολύ επιτυχημένη η αποστολή αυτή με επικεφαλή την Σεσίλ Κέγκε. Σεσίλ παρακαλώ. Για να μας πεις τι έγινε και ποια ήταν τα κυριότερα σημεία της επίσκεψής σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Κλόντ. Ήταν ε, μεγάλη ευχαρίστηση που ηγήθηκα της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου στο Φόρουμ των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το ΦΡΑ, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο Ο Φλάχτη, τον, ε, συγγνώμη, τον διευθυντή Ο για την παρουσία του σήμερα εδώ. Η παρουσία μας ε, κατέδειξε το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει η Επιτροπή μας για μια πιο ισχυρή σχέση θεσμική με τη μοναδική αυτή υπηρεσία που εγγυάται και επιτηρεί την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάτι που είναι γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Είδαμε απευθείας και συμμετείχαμε στις έξι ολομέλες και στις διάφορες ομάδες εργασίας. Ήρθαμε σε επαφή με τις κύριες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και συμβάλαμε στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων της ΦΡΑ μέχρι το 2022 όπως είπα σε πολλές από τις παρεμβάσεις μου, η Ένωση έκανε πολλά τις τελευταίες δεκαετίες για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλές διακρίσεις καταργήθηκαν. Πολλοί φραγμοί. Και επιτέλους είχαμε το πολιτικό θάρρος να ενεργοποιήσουμε τις διαδικασίες του άρθρου 7. Και τώρα έχουμε να επιτεθούμε σε άλλες μορφές διακρίσεων. Ευχαριστώ δημοσίως τον ε, Διευθυντή κύριο Φλάρτη που στήριξε τη μάχη μας, της Επιτροπής μας δηλαδή, για τα κυριότερα θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τον ευχαριστώ που εκφράστηκε υπέρ μια στρατηγικής κατά ε, της ε, ομοφοβίας. Επίσης, η δουλειά που κάναμε για την ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης ήταν ε, πολύ σημαντική. Με βάση τα στοιχεία σας μπορέσαμε να διαμορφώσουμε μία ε, στρατηγική για την ε, καταπολέμηση των διαχρήσεων κατά των προερχομένων από την Αφρική. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, χαίρομαι για την πλήρη διαθεσιμότητα και τις ιδιαίτερες ικανότητες όλων των συνεργατών σας. Πάντα ήταν πρόθυμοι να ικανοποιήσουν τα αιτήματά μας για όλα τα θέματα για όλες μας τις εργασίες. Πολλά έχετε κάνει, αλλά και πολλά ακόμη πρέπει να κάνετε. Ιδιαίτερα γιατί έχουμε νέες προκλήσεις που, που βλέπουμε στον ορίζοντα. Για παράδειγμα, αυτό το πολιτικό κλίμα μίσους και διακρίσεων που βλέπουμε στην Ευρώπη, που ενισχύεται από τις ε, λαϊκιστικές και ξενοφοβικές δυνάμεις. Όλα αυτά διακυβεύουν κάθε μέρα τις αξίες από τον οποίων βασίζεται η Ευρώπη μας. Εργαστήκαμε και για την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων που εφαρμόζεται. Είναι θέμα επιβίωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμογή της. Με τον εκτελεστικό διευθυντή συζητήσαμε και τα θέματα επί των οποίων πρέπει να επιμείνουμε περαιτέρω. Ιδιαίτερα παραβιάσεις των ε, δικαιωμάτων που έχουν να κάνουν με τα εγκλήματα μίσους, είτε διαδικτυακά είτε όχι, εκμετάλλευση των ε, ανηλίκων και η κατάσταση των ε, ε, μεταναστών που είναι μέχρι και σήμερα από την Πομπέη Τράγη, από τις, πολιτιστι... από τις ε, λαϊκιστικές ε, κυβερνήσεις οι οποίες ποινικοποιούν την ανθρωπιστική βοήθεια όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Ακουάριου και ενός άλλου σκάφους τώρα βλέπουμε τι γίνεται με το σκάφος Μάρε Ιόνιο Ιόνιο Πέλαγος δηλαδή και θα είδατε τη δήλωση ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών ο οποίος έκανε τέσσερα απαράδεκτε δηλώσει. Σα καλώ να το καταδικάσετε ανοιχτά. Ω ε, πρόεδρο αντιπροσωπεία είχα την ευχαρίστηση να συμμετάσχω στη συνεδρίαση τη ΦΕΜΠ, που είναι η ομάδα εργασία για ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Θεμελιώδη δικαιώματα. Και υπέγραψα, ε, τη σημασία τη δημιουργία ενό διαθρωμένου και τακτικού διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών. Και επέμεινα ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει ένα ρόλο. Μαζί με τη ΦΡΕΜΠ και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές των κρατών μελών για την ε, αξιολόγηση των ε, εθνικών νομοθεσιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάνω μία έκκληση. Δεν μπορούμε να ζητάμε από την ΦΡΑ να αντιμετωπίσει τις διάφορες προκλήσεις χωρίς να την προκοδοτήσουμε με τις επαρκείς πιστώσεις. Η ΦΡΑ πρέπει να διευρύνει το πεδίο λειτουργίας της, να ενισχύσει τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τα εθνικά κοινοβούλια για να διαμορφωθούν νέες στρατηγικές για να αντιμετωπιστεί αυτό το κλίμα μίσους και διακρίσεων που εξαπλώνεται στην Ευρώπη. Και για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να αυξήσουμε τους πόρους. Ευχαριστώ για μια φορά τον ε, Διευθυντή Οφλάερτη και όλους τους συνεργάτες του για την ε, υποδοχή που μας έκαναν στη Βιέννη. Ελπίζω να μπορέσω να συμμετάσχω, να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε και στο επόμενο φόρουμ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ σε για αυτή την παρουσίαση που καταδεικνύει, παρουσίαση, συγγνώμη, που καταδεικνύει πόσο περίπλοκη είναι η εργασία που έχει ενώπιον της τώρα η ΦΡΑ λόγω του πολιτικού κλίματος που υπάρχει. Γιατί πρέπει να εργαστεί για όλη την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο. Και όπως υπόθηκε κάνει ό,τι μπορεί. Ανταποκρίνεται στα μεμονωμένα αιτήματα των μελών. Κάτι που τόνισε και στο παρελθόν ο διευθυντή, Αλλά είναι κάτι δύσκολο. Τη μια μέρα πρέπει να ασχοληθεί με τη Μεσόγειο, την άλλη μέρα πρέπει να ασχοληθεί με την αφροφοβία. Όλα αυτά τα θέματα είναι πολύπλοκα. Ο Μάικλ τα έχει πει επανειλημμένα. Θα το πει και τώρα. Αλλά το φόρουμ ήταν πολύ καλή εκδήλωση. Είναι πολύ περίπλοκη η εργασία του, μην το ξεχνάμε. Και νομίζω ότι έχουν υπάρξει σημαντικέ επιτυχίε και σίγουρα βέβαια έχει και πολλέ προκλήσει ε, πάντα ενώπιον του. Μάικο, παρακαλώ, θα απαντήσει και μετά θα μιλήσουν και οι άλλοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου και τη δική σας και της κυρίας Κέγκε για τη σχέση που έχετε με την υπηρεσία σας. Μα για σας ε, εργαζόμεθα. Αυτό πάντα ήταν πρωταρχική προτεραιότητα για μας. Η στήριξη που δίνουμε στο Κοινοβούλιο για να στηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ενημερώσω τους συνεργάτες μου ότι, επιτύχουμε, ότι έχουμε επιτύχει είναι αποτέλεσμα της συλλογικής εργασίας 110 συνεργατών. Πολλά υπόθηκαν. Θα αναφερθώ σε ορισμένα. Εγώ είμαι ιδιαίτερα υπερήφανο για τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε για την αφροφοβία. Ξέρω πόσο συνέβαλε στη συζήτηση, ούτως ώστε να αποκτήσει περισσότερη σημασία το θέμα αυτό. Με ανησυχεί τώρα το φαινόμενο της Ισλαμοφοβίας. Και σε κάθε ευκαιρία το τονίζω. Ο φορέας μας σας έχει δώσει πολύ ενημερωμένα στοιχεία για ε, το πώς διαμορφώνονται και στα 28 κράτη-μέλη τα φαινόμενα Ισλαμοφοβίας. Τώρα για το φόρουμ. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Κέγκε και την αντιπροσωπή για τη συμμετοχή της και ευχαριστώ και εσάς Πρόεδρε που παίξατε βασικό ρόλο σε αυτό το φόρουμ. Αλλά και η Αντιπρόεδρος Μαγκίνες βοήθησε και άλλοι εδώ στο Κοινοβούλιο. Εκτιμάμε ιδιαίτερα το ρόλο που έπαιξαν, ε, έχει παίξει το Κοινοβούλιο για τι διάφορε δραστηριότητε του Φόρουμ. Και ορίζω Διάβασαν πολύ ενδιαφέρον το σχέδιο έκθεσης. Πολύ αναλυτικά αναφέρεται στην πόση ενέργεια υπήρξε σε αυτό το φόρουμ που είναι η τακτική κύρια εκδήλωσή μας η εμβληματική μας εκδήλωση εκεί συμμετέχουν διαφορετικές ομάδες και συζητούν τις κοινέ του ανησυχίε για τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση. Δεν έχω χρόνο για να σας μιλήσω για όλες τις ομάδες. Αν ναι, είναι όλες οι προφανείς ομάδες και μετά κάποια όχι τόσο συνήθιοι, όπου ασχολούμεθα με νέα θέματα. Αναφερθήκατε στο ΦΡΕΜΠ και θα αναφέρω και το ΚΟΧΟΜ, άλλο σημαντικός ε, χώρος εργασίας. Είχαμε 700 συμμετέχοντες και μας είπαν ότι ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων, αλληλοστήριξης. Αλλά όλα αυτά μετά πρέπει να έχουν και επιπτώσεις ε, στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και έχουμε ένα έγγραφο που λέγεται δήλωση του Προέδρου και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτά που ε, περιέχονται σε αυτό το έγγραφο. Για παράδειγμα, Όπω είπε η κυρία Κέγκε, εστιάσαμε κυρίω στο πώς να αξιοποιήσουμε καλύτερα την χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, στις δημόσιες συζητήσει στην Ένωση. Προέκυψαν πολλές ιδέες που τώρα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τώρα που είναι επέτειο της χάρτας. Για παράδειγμα, να υπάρχουν στοιχεία με δεδομένα αναχώρα. η πλευρά θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, του κράτους δικαίου. Και αυτό το συζητήσαμε. Και ε, στα απορίσματα της Προεδρίας αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα. Μετά το διάλογο του Συμβουλίου για το κράτος δικαίου. Και τα παιδιά των μεταναστών, για παράδειγμα. Εστιάσαμε ιδιαίτερα στα θέματα των παιδιών, που είναι τμήμα της ε, συζήτησης για το μεταναστευτικό. Έτσι νομίζω ότι εστιάζουμε το ενδιαφέρον για τα παιδιά για όλα τα μεταναστευτικά θέματα. Τώρα, σύντομα για το μέλλον. Πώς θα δημοσιεύει το φόρουμ στο μέλλον. Είχαμε μια εξωτερική αξιολόγηση του φόρουμ. Έχουμε τα απορίσματα, θα τα συζητήσουμε το Μάιο για να δούμε πού θα πάμε στο μέλλον. Δεν μπορώ να προκαταλάβω αυτή τη συζήτηση. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχιστούν αυτά τα περιοδικά φόρουμ και θα προτείνω στο Διοικητικό μου Συμβούλιο ότι το επόμενο φόρουμ πρέπει να γίνει το 2020. Σας ευχαριστώ πολύ για το έντονο ενδιαφέρον σας και για την ευρεία και ζωηρή συμμετοχή σας. Ευχαριστώ. Θα μπορούσαμε να φέρουμε πολλά άλλα θέματα. Αλλά ευχαριστώ που εστιάσατε στο φόρουμ, που νομίζω ότι ήταν πολύ επιτυχές. Οπότε, ο Τόμας Ζεντόφσκι επίσης συμμετείχε. Μόλις ήρθε. Τόμας. Να μας πεις κι εσύ. Ευχαριστώ πολύ, Μάικλ, για τη συμμετοχή σου. Ευχαριστώ, Κλοντ, που μου έδωσε το λόγο. Η συνεργασία μας με την ΦΡΑ είναι μία από τις καλύτερες συνεργασίες που έχουμε. Την επισκέφθηκα παρελειμμένα και υπό τον προηγούμενο διευθυντή και πρέπει να πω είναι πραγματικά άψογη. Εγώ που είμαι ο μόνιμος σκιώδης από πλευράς ΕΛΚΑ έπρεπε να αναφέρω μία υπηρεσία που πάντα τα πάει καλά και δεν δημιουργεί προβλήματα θα ανέφερα οπωσδήποτε τη ΦΡΑ είτε πρώτη είτε πρώτη δεύτερη. Πολύ σημαντική εργασία της. Ορισμένοι μπορούν να θεωρούν σήμερα ότι μια υπηρεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορούσε να έχει ίδια προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά εσείς δεν έχετε. Άρα δεν μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί τον οργανισμό σας, την υπηρεσία σας για να επικρίνει την Ένωση. Και αυτό εν ώψη εκλογών εμείς, τα κράτη της Κεντρικής Ευρώπης, είμαστε ιδιαίτερα εκτεθειμένα στην ρωσική προπαγάνδα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί αυτό. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η εργασία σας είναι πραγματικά άμομη και έχουμε συμμετάσχει στα φόρουμ αυτά. Εντάξει, αυτά που λέγονται μπορούν να ερμηνευτούν με διάφορα να εξεταστούν από διάφορε οπτικέ γωνίε. Εγώ γενικά έχω συντηρητικέ απόψει. Αλλά άλλοι έχουν άλλε. Και το βασικό είναι να μπορούν να κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και να κάνουν σοβαρέ συζητήσει. Νομίζω ότι αυτά δίνουν, δίνουν μια νέα διάσταση στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Οποτεδήποτε σας έχω ζητήσει ε, να μου αποστείλετε κάποια στοιχεία, μέσα σε μια εβδομάδα το πολύ μου τα έχετε στείλει και αυτό είναι ευχάριστη έκπληξη. Και αυτά που κάνετε γενικά η εργασία σας, μετανάστευση για παράδειγμα, ε, διακίνηση παιδιών, η κακοποίηση παιδιών. Πάντα μας δίνετε τα στοιχεία όταν τα ζητάμε. Πρέπει λοιπόν να σας στηρίξουμε, οπωσδήποτε. Μακροπρόθεσμα. Τώρα, ένα θέμα που δεν έχει να κάνει τόσο απευθεία με ε, τη δουλειά σα. Μήπως θα πρέπει να δείτε και τη διάσταση του φίλου, διαρωτώ με. Γιατί είναι μικρός ο φορέας σας. Έχει έννοια να επιχειρείτε ως τόσο μικρός φορέας να κάνετε τόσα πράγματα. Μπορεί ένας ε, τόσο μικρός φορέας να τα κάνει όλα ή πρέπει να είστε τμήμα ενός μεγαλύτερου φορέα γιατί μέχρι στιγμής είναι άριστες εκθέσεις σας, άριστες πραγματικά κυριολεκτό. Ποτέ δεν έχω διαβάσει έκθεση δική σας. που να μου φαίνεται βελτιώσιμη. Και η ποιότητα, ξέρετε, της εργασίας μας εδώ στη ΛΥΜΠΕ σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στη δική σας τη δουλειά. Βεβαίω έχουμε συμβιωτική σχέση, πρέπει να αλληλοστηριζόμεθα. Αυτό είναι σαφέ. Η έκθεση της Σεσίλ Κιέγγε αναφέρεται σε όλου του τομεί ε, αρμοδιότητά σας και ουσιοδό. Και νομίζω ότι συμφωνούμε σχεδόν σε όλα. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε αυτή τη δυνατότητα σήμερα να εδραιώσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με βάση και την αποστολή αυτή και ελπίζω και η επόμενη θητεία θα συνεχίσει να συνεργάζεται πολύ καλά όπως και εμείς την τελευταία πενταετία. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Σπινέλη. Εγώ συμφωνώ με τις ευχαριστίες του Πρόεδρου μας προς το πρόσωπο του κυρίου Φλάχερτη και ευχαριστώ ιδίως τον οργανισμό σας για την ε, στενή και ενεργό συνεργασία ήδη από τότε που συνεργαστήκατε με την Επιτροπή Συνταγματικών για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και εκεί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η διερεύνηση των υποχρεώσεων του Οργανισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνεργασία αυτή μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Έχω μία ερώτηση. Η έκθεση που δημοσιεύτηκε για την εφαρμογή των διατάξεων του χάρτη ζητεί συστηματική συμμετοχή στις νομοθετικές εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό για μένα είναι και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ως εισηγήτρια για το θέμα αυτό, κάτι που διαφεύγει δηλαδή των ορίων αρμοδιότητας του φόρουμ γιατί θα πρέπει όπως είπα να γίνει με τρόπο συστηματικό και εκεί βρίσκω ότι υπάρχει δυσκολία διότι τι σημαίνει αυτό και πώς μπορεί να οργανωθεί μια τέτοια συνεργασία για μένα δεν είναι πολύ σαφές αυτό δεν διατυπώνεται σαφώς την έκθεση ε, δηλαδή γύρεται η αξίωση αυτή αλλά θα ήθελα να μάθω πώς θα εφαρμοστεί και ποια θα ήταν η καλύτερη αντίδραση απέναντι σε αυτή την αξίωση. Ευχαριστώ Μπάρμπαρα. Άλλος κανείς? Όχι. Μάκελος, εσείς ορίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ και τα μέλη σας για τις ε, πολύ ευγενείς παρατηρήσεις τις οποίες θα μεταφέρω στους συναδέλφους στην Βιέννη. Ευχαριστώ τον κύριο Ζεχόφσκι για τη συμμετοχή του στην αποστολή αλλά και τις ερωτήσεις. Εξετίμησα ιδιαίτερος το γεγονός ότι ευχαριστείτε για το έργο του οργανισμού μας και για την ποιότητα του και για την ταχύτητα. Η ταχύτητα είναι σημαντική για σας, αλλά και η ποιότητα επίσης για να γνωρίζετε ότι μπορείτε να βασίζετε σε εμάς και ασφαλώς θα συνεχίσουμε να φροντίζουμε τα δύο αυτά στοιχεία. Για το ζήτημα των φύλων υπάρχουν ίσως δύο θέματα εδώ. Αφενός να περιλάβουμε το θέμα αυτό σε οτιδήποτε κάνουμε και επίσης ένας οργανισμός που στοχεύει ιδιαίτερα στα θέματα ισότητας των φύλων. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, σας βεβαιώ ότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ισότητα των φύλων σε όλα, στο μεταναστευτικό, ε, τις διαφορετικές ε, εμπειρίες ανδρών και γυναικών. Αυτά παραμένουν πολύ σημαντικά για μας. Σε ό,τι αφορά τώρα τον πρωταρχικό στόχο για την ε, ισότητα, ε, υπάρχει και άλλος οργανισμός που είναι αυτός που είναι ο αδελφός οργανισμός δηλαδή. Δεν θα κάνω όλες τις παρατηρήσεις σχετικά. Ευχαριστώ και την κυρία Σπινέλη για τα ευγενικά της λόγια. Πολύ ευχαρίστως δημοσίευσαμε τη γνωμοδότηση για τον χάρτη ε, στην προπαρασκευή της της επαιτίου και υπάρχει και εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης χθε και σήμερα ώστε να αρχίσουμε με κάποιο κάποιο πιο επίσημο τρόπο την, ε, τον εορτασμό της επαιτίου αυτής για την χρήση του χάρτη από όλε τις ενδιαφερόμενες ομάδες για το ειδικότερο ερώτημα της κυρίας Σπινέλη σχετικά με το ρόλο του οργανισμού στο νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό να αρχίσω λέγοντας ότι ήδη παίζουμε σημαντικό ρόλο με την παραγωγή δεδομένων. Δηλαδή σας προσφέρουμε τα δεδομένα, τα στοιχεία που χρειάζεται για να κάνετε τις αναγκαίες επιλογές. Και αυτό είναι ο πυρήνας του έργου μας και θα συνεχίσει να είναι. Και καθώς και έρευνε. Οι έρευνε, η ποιότητα της ερευνητικής εργασίας που σας μεταφέρουν τις φωνές των δικαιούχων και θα συνεχίσουμε να το φροντίζουμε ιδιαίτερα αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα συγκεκριμένες νομοδοτήσεις για ε, νομοσχέδια, εκεί μας περιορίζει ο κανονισμός μας και μπορούμε να το κάνουμε μόνο εφόσον λάβουμε αίτηση από εσά. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνεται πάντοτε στην βάση ad hoc request, δηλαδή εφόσον μας ζητείτε κάτι συγκεκριμένα. Και θα εξαρτηθεί αυτό και από την ε, ε, αρμοδιότητα που έχουμε στον τομέα αυτό, αλλά και από την, ε, τις ικανότητες που θα διαθέτουμε, δηλαδή αν θα έχουμε το αναγκαίο προσωπικό και μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ Μάικλ. Νομίζω ότι εκμεταλλευτήκαμε καλά την παρουσία σας σήμερα εδώ και ας προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. ανταλλαγή απόψεων για το φαινόμενο του αντισημιτισμού στην Ευρώπη που έχουν ζητήσει οι συντονιστές. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκε στο φόρουμ του οργανισμού σας και θελήσαμε να το βάλουμε ωστόσο συγκεκριμένα στην ημερήσια διάταξη. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στη συζήτηση αυτή τώρα. Σας ευχαριστώ και πάλι που ε, είχατε τη διάθεση να κάνετε τη σχετική εισαγωγή για θέματα αντισημιτισμού στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που έθεσε το ζήτημα του αντισημιτισμού στην Μερσια Διάταξη και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σντεχόφσκι που ηγήθηκε ε, το προσπάθειας αυτής. Ε, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ, εμένα να σας πω ότι υπάρχει πρόβλημα ε, αντισημιτισμού στην Ευρώπη είναι πονίδιστο ε, και δυστυχώς το πρόβλημα είναι μεγάλο. Πριν πέντε χρόνια που κάναμε μία μελέτη είδαμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με μεγάλες διαστάσεις και πέρυσι το Δεκέμβριο δημοσιοποιήσαμε εκ νέου την έρευνα, την οποία επαναλάβαμε ε, και ήταν μεγαλύτερη με 16.000 απαντώντες ε, από 12 κράτη-μέλη ε, εβραϊκής καταγωγής. Δεν είναι όμως το θέμα ότι είναι μόνο από 12 χώρες. Μιλάμε για Εβραίους από όλη την Ευρώπη ουσιαστικά. ακούσαμε φωνές που εκπροσωπούν το 96% της εβραϊκής κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειλικρινά τα αποτελέσματα ήταν άκρο ανησυχητικά. Θα σας δώσω ορισμένα στοιχεία. Το 85% ε, των ε, Εβραίων ε, έτσι προσδιορίζονται οι ίδιοι έτσι, ως Εβραίοι. Το 85% είπα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή τους δεν είναι ούτε η ανεργία, ούτε η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη ή κάποιο άλλο σχετικό ζήτημα, αλλά ο αντισημιτισμός. Το 85% το είπε. Το 90% των απαντώντων μας είπαν ότι έχει αυξηθεί το φαινόμενο του αντισημιτισμού τα τελευταία πέντε χρόνια. Το 1% λένε ότι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα στο διαδίκτυο. Το 73% στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, το 71% στα μίντια και το 70% στην πολιτική. σε ό,τι αφορά προσωπική παρενόχληση, το 1 τρίτο περίπου, το 28% είπαν ότι έχουν ε, υποστεί ε, ε, παρενόχληση το τελευταίο έτος προσωπικά οι ίδιοι και αν φορούσαν την ιδιαίτερη χαρακτηριστική τους ενδυμασία ήταν ακόμα περισσότερες οι πιθανότητες να υποστούν κάποια επίθεση. Ε, λέμε ότι οι γυναίκες έχουν ε, πιο δυσάριστες εμπειρίες ε, συνήθως σε ό,τι αφορά την παρενόχληση, αλλά εδώ η χαρακτηριστική ενδυμασία είναι αντρική κυρίως, οπότε οι άντρες το έχουν αντιμετωπίσει. 40% φοβούνται ότι θα τους επιτεθεί κάποιος. Και αυτό με φέρνει σαν από τα πιο ανησυχητικά ε, νούμερα ότι το 38% λόγω φόβου λένε ότι έχουν σκεφτεί να μεταναστεύσουν. Αυτό πραγματικά ε, εμένα μου δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Φαίνεται ένα μεγάλο ποσοστό να θέλει να φύγει για να αναστήσει ασφάλεια. Το 80% επίσης δεν αναφέρουν ε, τα περιστατικά και είναι σημαντικό το νούμερο αυτό. Γιατί λέει ότι ό,τι ο επίσημο στοιχείο έχουμε ε, είναι πραγματικά πολύ χαμηλότερο σε σχέση με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και 70% των απαντώντων εκφράζουν την άποψη ότι δεν κάνουν αρκετά τα κράτη για να εξασφαλίσουν την προστασία τους και την ασφαλεία τους. Και ολοκληρώνω τις στατιστικές αυτές αναφορές ε, σε ένα στοιχείο από το Ευρωβαρόμετρο του Ιανουαρίου. Από την Κομισιόν δηλαδή που λέει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο 43% λένε ότι δεν είναι και μεγάλο θέμα ο αντισημιτισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μισό δηλαδή του γενικού πληθυσμού δεν βλέπει πρόβλημα ενώ σχεδόν όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το αντιμετωπίζουν ως ένα σοβαρό πρόβλημα, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τι να κάνουμε λοιπόν με αυτό. Αρχικά πρέπει να αναγνωρίσουμε πόσα ήδη γίνονται. Εσείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγκρίνατε ένα πολύ σημαντικό ψήφισμα για την ε, καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε μια πολύ αξιέπαινη πρωτοβουλία, διόρισε συντονιστή για θέματα αντισημιτισμού. Η ομάδα υψηλού επίπεδου για την αντιμετώπιση ρατσισμού, ξενοφοβία και άλλων μορφών μυσαλλοδοξία επίση κάνει πολύ σημαντικό έργο, στηρίζοντα ε, την καταγραφή και δίωξη τέτοιου είδου εγκλημάτων μίσου. Και βέβαια πάρα πολύ μεγάλη είναι και η σημασία τη διακήρυξη διακήρυξης που ενέκρινε το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2018. Σε σχέση με τη δήλωση αυτή, έγιναν σημαντικές αναγγελίες από την Επίτροπο Γιούροβα πριν από λίγες εβδομάδες και τέλος, ε, στα πλαίσια πάντα αυτή της ε, έναρξης δράσης, ε, της αφετηρίας, Εκτιμώ ιδιαίτερα και το έργο της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τη μνήμη του Ολοκαυτώματος. Προεδρεύει το Λουξεμβούργο αυτή τη στιγμή αυτής της συμμαχίας που έχει και έναν ορισμό πάρα πολύ χρήσιμο που μας καθοδηγεί στο δικό μας έργο αλλά και άλλους βέβαια φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε λοιπόν να ε, θεωρήσουμε ότι έχουμε μια πολύ καλή βάση και να αντλήσουμε από αυτήν. Έρχομαι σε κάποιες συστάσεις. Πρώτα απ' όλα από το έργο μας ε, και μας το λένε και οι εβραϊκές αυτές ομάδες και ενώσεις. Πρέπει η δουλειά να γίνει όχι για, αλλά μαζί με τους Εβραίους. Συνεργασία δηλαδή για να προσδιοριστούν οι προκλήσεις και να αντιμετωπιστούν. Δεύτερον, οι νέε πρωτοβουλίε για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού πρέπει να εστιάσουν στην εκπαίδευση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι επιζώντε του ολοκαυτώματο ε, πεθαίνουν, χάνονται και σε αυτούς βασιζόμασταν για να πούν την ιστορία τους στις νέες γενιές. Από εδώ και πέρα αυτό δεν θα είναι δυνατό. Πρέπει να βρούμε νέους τρόπους για να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας και να τους μάθουμε ε, τη φρίκη του ολοκαυτώματος για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Τρίτον, και τα λέω έτσι πολύ πεζά, πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά για να εξασφαλίσουμε τη σωματική προστασία ε, και των ανθρώπων και την ηλική προστασία των εγκαταστάσεων, δωρεάν προστασία. Το ότι θα πρέπει να πληρώνουν οι εβραϊκές ομάδες για την προστασία τους είναι μεγάλο πρόβλημα. Και τέλος, να καταπολεμήσουμε καλύτερα τον αντισημιτισμό με μεγαλύτερη ε, καλύτερη εφαρμογή της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη. Και υπάρχουν νομοθετήματα για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Επίσης, είπα τέλος, αλλά έχω και κάτι ακόμη να πω. Η καταπολέμηση του αντισημιτισμού βέβαια, ότι θα παραμείνει ε, στο επίκεντρο της ταυτότητας ε, και των αρμοδιοτήτων του οργανισμού μας. Θα κάνουμε συνεχώς έρευνες και σε εθνικό επίπεδο. Περιοδικά ε, θα επαναλάβουμε αυτή την πανευρωπαϊκή έρευνα. Ήδη έχουμε ετήσια επικαιροποίηση των στοιχείων που συλλέγουμε για τον αντισημιτισμό στην Ευρώπη. Βέβαια, πρέπει να έχετε υπόψη ότι η ποιότητα των δεδομένων είναι ανομοιόμορφη, ανομοιογενής. Επίση, ό,τι αφορά τη μνήμη του ολοκαυτώματο, στηρίζουμε τι σχετικέ πρωτοβουλίε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ένωση, την Κομισιόν, στον ηγετικό ρόλο που έχουν για την μάχη αυτή, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, που έχει να δώσει η Ένωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, Μάικλ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Στεχόφσκι, στην κυρία Σπινέλη και στον κύριο Κέστερ. Κύριο Στεχόφσκι. Ευχαριστώ, Κλοντ. Ευχαριστώ τον Μάικλ για τις απαντήσεις του και για το γεγονός ότι καταφέραμε να διοργανώσουμε αυτή τη συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω του συντονιστέ λοιπόν από όλε τι πολιτικέ ομάδε που συμφώνησαν με τη σύστασή μου να συζητηθεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως αντισημιτισμό πριν τη λήξη τη κοινοβουλευτική θητεία. Πιστεύω πως η παρουσίασή σας εδώ ένα πράγμα καθιστά ξεκάθαρο ότι το μίσος, ο αντισημιτισμός, το μίσος ε, κατά των Εβραίων εξαπλώνεται, εξαπλώνεται όλο και περισσότερο, όλο και μακρύτερα. Ε, συνάντησα εκπροσώπους των εβραϊκών κοινοτήτων διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών και πρέπει να σας πω ότι ήδη από το 2015 τα κράτη-μέλη μας προειδοποιούν συστηματικώς για φραστικές επιθέσεις σε βάρος Εβραίων, αλλά κάτι ακόμη χειρότερο, σε όλο και περισσότερα κρούσματα ε, σωματικής βίας ε, και επίθεσης. Πριν ένα χρόνο ήμουν στη Σουηδία και εκεί ήδη έχει αναφερθεί το Μάλμο, αλλά ε, Τέτοια είναι η κατάσταση που γονεί αναγκάζονται να ε, πάρουν τα παιδιά του από το σχολείο για να μην δεχτούν επιθέσει. Ερωτώ λοιπόν, γιατί αφού είναι η Σουηδία πλούσια και ευημερούσα χώρα και αυτό ε, το πηγαίνω και συνολικά στην Ευρώπη. Αφού υπάρχει ευημερία, υπάρχει πλητός γιατί ο αντισημιτισμός. Ξεχάσαμε την ιστορία, ξεχάσαμε τη φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης. και στο δημόσιο διάλογο που γίνεται. Δεν υπάρχουν τόσοι που γράφουν ε, ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό που αρχίσαμε και νομίζω πρέπει να ασκηθεί πίεση σε πλατφόρμες ώστε να μην παίρνουν τέτοιου είδους αντισημιτικά σχόλια. Να καταπολεμήσουμε αυτόν τον εξτρεμισμό και όταν παραβιάζονται οι κανόνες του δημοσίου διαλόγου, όταν κανείς ε, δείχνει ακραία δείγματα επανειλημμένως πρέπει να διαγράφεται, να αποκλείεται από το κοινωνικό διάλογο. Αυτό πρέπει να το φροντίσουν διάφορες πλατφόρμες. Το ερώτημά μου είναι γιατί το Ισραήλ που θέλει να είναι το μοντέλο της σύγχρονης δημοκρατίας ε, προχωρεί σε νέους επικισμούς για δεκάδες χιλιάδες Εβραίους που θα μεταβούν εκεί από τη Γαλλία. Γιατί φτιάχνει επικισμούς για Γάλλους Εβραίους το Ισραήλ. Γιατί αυξάνεται η εβραϊκή κοινότητα στην Αμερική, ε, κυρίως Γερμανοί. Και υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστώ το φαινόμενο του Μπορούν τα κράτη-μέλη αρκεί να εφαρμόσουν σωστά την νομοθεσία και τους κανόνες. Είναι απαράδεκτο και το έχω ξαναπεί αυτό που συμβαίνει σε ορισμένα κράτη-μέλη σήμερα. Είναι απαράδεκτο. Πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά του, Να εκθέσουμε το πρόβλημα. Γιατί αν χάσουμε τη μάχη κατά του αντισημιτισμού, θα χάσουμε και τον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ, Ιμπάρο. Ευχαριστώ, Κλοντ. Και εγώ συμμερίζομαι την ανησυχία και το φόβο που έχω έναντι της αύξησης του αντισημιτισμού. Δύο ερωτήσει. Αναφερθήκατε σε διάφορα ποσοστά για το πόσοι Εβραίοι θέλουν να φύγουν από τις χώρες της Ένωσης. Ε, μήπως έχετε στοιχεία για το πού θέλουν να πάνε αυτοί που θέλουν να φύγουν. Για παράδειγμα. Εγώ ε, ε, που αν ήμουν Εβραία εάν ήθελα να φύγω από την Ευρώπη δεν θα ήξερα που να πάω. Και το δεύτερο τον ορισμό του αντισημιτισμού. Ξέρετε πολύ καλά ότι το επιχείρημα αυτό ε, αμφισβητείται ιδιαίτερα και μεταξύ των Εβραίων. Το επιχείρημα του πώς ακριβώς ε, ορίζει αυτή η συμμαχία κατά για την ε, μνήμη του ολοκαυτώματος την, τον αντισημιτισμό. Διότι ορισμένοι Εβραίοι λένε ότι, αυτό, ορισμένοι λένε ότι το γεγονό ότι περιλαμβάνει και την επίκριση κατά τη πολιτική του κράτου του Ισραήλ, του κράτους του Ισραήλ είναι ε, προβληματικό. Επίσης, ο οργανισμός σας ποτέ δεν έχει υιοθετήσει αυτόν τον ορισμό της συμμαχίας. Πρόκειται να τον ε, ε, υιοθετήσετε, μήπως τον έχετε πρόσφατα υιοθετήσει ή θα εξακολουθήσετε να επιμένετε ότι είναι καλύτερα ο οργανισμός σας να μην υιοθετήσει αυτόν τον ορισμό του αντισημιτισμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μπάρμπαρα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Κώσταρ. Ευχαριστώ Κλοντ. Ευχαριστώ για την έκθεσή σας, την παρουσίασή σας. Χαίρομαι που είπατε ότι βασικό καθήκον σας θεωρείτε ότι είναι ακριβώς η καταπολέμηση του αντισημιτισμού, κάτι που πραγματικά είναι έγνοια σας. Και είπατε, σαφώς, κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι ιδιαίτερα λυπηρό. Μετά το ΣΟΑ, 38% των Εβραίων μελετούν το ενδεχόμενο να φύγουν από την Ένωση και από την άλλη μεριά 50% των πολιτών της Ένωσης δεν θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα αντισημιτισμού εδώ, υπάρχει μεγάλη αντιστοιχία και μεγάλη ανάγκη να δράσουμε. Γιατί όμως, γιατί και πώς είναι δυνατόν τόσοι Εβραίοι συμπολίτε μας, άνδρες και γυναίκες, να αισθάνονται ότι απειλούνται σε τέτοιο βαθμό, διότι, εδώ μεταξύ, κυβερνήσεις ε, που ελέγχονται από ακροδεξιούς ε, λαϊκιστές προωθούν τον αντισημιτισμό. Για παράδειγμα στην Αυστρία είχαμε μια περίπτωση πρόσφατα όπου στο αυστριακό ραδιόφωνο κάποιος επενέθηκε ως πατριώτης και δημοκράτης ενώ είναι ανοιχτά ζει και αντισημίτης. Και στην Ουγγαρία έχουμε τον ε, κύριο Όρμπαν, ο οποίος ε, κάνει εκστρατείε ε, με αντισημιτικά στοιχεία κατά της Ένωσης. Και στην Πολωνία, όπου η κυβέρνηση είναι στην πορεία έγκρισης ενός νομοσχεδίου που θα αμνηστεύσει τους Πολωνούς πολίτες για αντικείμενα που διαπράχθηκαν ε, κατά την περίοδο ΣΟΑ. Πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο που ορισμένοι προωθούν τον αντισημιτισμό. Και κάτι ακόμη. Πολύ συχνά υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ αντισιονισμού και αντισημιτισμού. Έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση για τον αντισιονισμό πολύ συχνά είναι πρόσχημα για να προωθηθούν ε, αντισημιτικές προκαταλήψεις. Μήπως μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό και επιπλέον. Τον ορισμό αυτό τον ορισμό αυτό της Διεθνούς Συμμαχίας ε, τον θεωρώ πολύ σωστό και πρέπει να παραμείνει. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω κι εγώ, Μάικο, Ξέρω ότι το έχει σκεφτεί. Το θέμα του ακροδεξιού εξτρεμισμού και της θεωρίας συνωμοσίας. Το έχετε εξετάσει. Ξέρω ότι έχετε δει τη σχέση του εξτρεμιστικού περιεχομένου με τις ε, εκδηλώσεις ακραίας βίας. Το πώς συνδυάζεται αυτό με αντισημιτικές ε, απόπειρες. Ξέρω ότι είναι περίπλοκο. Να δείτε κατά πόσο συγκλίνουν αυτά τα δύο φαινόμενα. Και αν θεωρείτε ότι τα αντισημιτικά επιχειρήματα... Αυτό για τη μεγάλη αντικατάσταση και τα αντιμεταναστευτικά μηνύματα θεωρείτε ότι συνδέονται με αυτή την ε, προπαγάνδα της ακροδεξιάς και συνδέονται και με τον αντισημιτισμό. Πώς αναλύετε το φαινόμενο αυτό. Συνδυάζονται αυτά τα φαινόμενα ή είναι διακριτά. Συμμετέχουν στην ε, ε, αύξηση του αντισημιτισμού στο ίντερνετ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ορισμένες ε, ερωτήσεις ε, στην ουσία επικαλύπτονται, οπότε δεν θα απαντήσω σε κάθε συγκεκριμένο. Θα συνδυάσω την απάντησή μου. Νομίζω ότι απαντώντας σχεδόν σε όλους θα έλεγα ότι θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτό το θέμα μόνο εάν καταλάβουμε σε τι βαθμό πρέπει να είναι πρωταρχική προτεραιότητα. Δεν μπορεί να είναι ένα μεταξύ των άλλων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι καθοριστική σημασία θέμα για την Ευρώπη. Μα για ποιο λόγο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν μπορεί να προστατεύσει τι εβραϊκέ κοινότητέ τη. Είναι τόσο αποτελεσματικό. Αν δεν τι προστατεύσει αποτελεσματικά, αποτυγχάνει συνολικά. Και σίγουρα και εγώ δεν θα ήθελα να ζω σε ένα τέτοιο μέρο. Και η προτεραιότητα σημαίνει ότι θα υπάρχει και επαρκή χρηματοδότηση και προσοχή. Εντό τη Ένωση Βλέπω όλο και περισσότερα στοιχεία ότι όντω ε, εστιάζουμε εδώ έχουμε την δήλωση του Συμβουλίου, τι πρωτοβουλίε τη ε, Επιτρόπου Γιούροβα για παράδειγμα. Και είναι μόνο δύο παραδείγματα. Τώρα, τι προκαλεί αυτή την άνοδο του αντισημιτισμού και πώ θα τον αντιμετωπίσουμε. Τώρα, από το ευρύτερο στο στενότερο. Το ευρύτερο που έχει να κάνει και με αυτό που είπατε εσεί, Πρόεδρε. Αναμφίβολα αυτό το ρεύμα λαϊκισμού περιέχει και ισχυρά στοιχεία συγγνώμη, αυτό το ρεύμα λαϊκισμού περιέχει ισχυρά στοιχεία, ισχυρά στοιχεία αντισημιτισμού, αναμφίβολο. Και τα ελεγιστικά μηνύματα βεβαίω περνάνε και από το διαδίκτυο. Οπότε πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και εκεί, τα αντισημιτικά. Αναφέρεσταν, ανα, συζητούσα όταν μπήκα σε μια μελέτη και είδα τι υπόθηκε εκεί ότι πρέπει να απαλήφονται τα ε, post μίσου χωρίς όμως να θίξετε την ελευθερία έκφρασης δεν θέλω να πάνε σε αυτή τη συζήτηση αλλά η υπηρεσία μου προσπαθεί να στηρίξει με κάθε τρόπο τη συζήτηση για το θέμα αυτό για παράδειγμα εστιάζουμε στην καλύτερη κατανόηση του τι ρόλο παίζει η τεχνητή νοημοσύνη και τι όρια πρέπει να τεθούν. στην ε, εφαρμογή της. Και δεν είναι άσχετο με αυτά που λέμε. Πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί για να σταματήσουμε για παράδειγμα τους κακόβουλους αλγόριθμους τώρα πιο στενά στον αντισημιτισμό. Σίγουρα Πρέπει να ενισχυθεί το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Δεν φταίει ο μισός πληθυσμός της Ένωσης που δεν θεωρεί ότι είναι θέμα ο αντισημιτισμός. Εμείς που έχουμε την ευθύνη ευαισθητοποίησης φταίμε στις ε, σχολικές αίθουσες αλλά και μεταξύ των ενηλίκων. Χρειαζόμαστε πιο μεγαλύτερη δημιουργικότητα, μεγαλύτερη φαντασία για το πώς να περάσει το μήνυμα. Τώρα, δεν ε, διώκεται και επαρκώς η αντισημιτική προπαγάνδα. Δεν τους ενθαρρύνουμε να κάνουν καταγγελίες και μηνύσεις. Οι περισσότεροι οι οποίοι είναι θύματα τέτοιων ε, ενεργειών δεν το αναφέρουν, αλλά πρέπει να πιστούν με σεβασμό, να το γνωρίζουν αυτό όταν θα τα καταγγείλουν αυτά τα πράγματα. Και κατόπιν πρέπει να γίνει μία σωστή ανάκριση και δίωξη. Μόνο όταν θα μπουν στη στενή ορισμένοι θα καταλάβουν και θα αλλάξει η κατάσταση. Για τον ορισμό τώρα αυτής της συμμαχίας η κυρία Σπινέλη αναφέρθηκε στην προϊστορία του ορισμού αυτού στις ε, προκάτοχες οργανώσεις. Εμείς δεν θεωρούμε ότι η δουλειά μας είναι να εγκρίνουμε ορισμούς. Οι ορισμοί είναι περισσότερο νομοθετικό θέμα θέτουν ε, το πλαίσιο και τις παραμέτρους εφαρμογής του δικαίου. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι αρμοδιότητά μας. Εμείς θέλουμε να σας στηρίξουμε για να εφαρμόζεται ο νόμος για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν καθορίζουμε τις παραμέτρους. Εμείς ε, δεν έχουμε το ίδιο ε, τις ίδιες αρμοδιότητες με τους προκατόχους και οι προκάτοχοί μας δεν είχαν υιοθετήσει τον ορισμό. Η συμμαχία αυτοί όμω, κατά του αντισημιτισμού, ενέκριναν ορισμό τον οποίο έχουν εγκρίνει οι θεσμοί τη Ένωση. Και μα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτόν τον ορισμό. Χρειαζόμαστε αυτέ τι παραμέτρου για να κάνουμε τη δουλειά μα και τώρα μα έχουν δοθεί και έτσι τι αξιοποιούμε. Αλλά εμεί δεν εγκρίνουμε ούτε επικυρώνουμε ορισμού, δεν είναι δουλειά μα. Τέλο. Ποιοι επιθυμούν να μεταναστεύσουν και πού. Θα σας στείλω αναλυτική απάντηση. Αλλά από ό,τι ξέρω τώρα, στι περισσότερε περιπτώσει λένε ότι θέλουν να πάνε στο Ισραήλ. Αλλά μ, υπάρχουν και άλλοι που θέλουν να πάνε αλλού. Θα σα δώσω πιο αναλυτικά στοιχεία αργότερα και ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι, και εμένα, Μπάρμπαρα, πολλέ φορέ όταν με βλέπουν μου λένε γύρνα πίσω στην Ινδία. Το παθαίνω. Τέλο πάντων. Δεν βλέπω να σας διασκέδασε αυτό που είπα. Λοιπόν, αυτό που καταδεικνύει πόσο διαφορετική είναι η τομή ε, αρμοδιότητά σας, να περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η γνωμοδότηση για τα hotspot στην Ελλάδα και την Ιταλία. Όταν ξεκινήσατε τη δουλειά σα για τον οργανισμό αυτό, ξέρω πόσο λίγο προσωπικό είχατε. Γιατί είναι περίπλοκη δουλειά, πρέπει να γίνει επιτόπου αλλά και πάλι νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμα αυτά που μας στείλατε όπως και όλα τα άλλα στοιχεία που μας στείλατε για πολλά θέματα γιατί φαίνεται και γι' αυτό να έχουμε την άποψη του οργανισμού σας για το τι γίνεται στην Ελλάδα και την Ιταλία είναι σημαντικό για αυτή την γνωμοδότηση του περασμένου Φεβρουαρίου. Μάικρο, παρακαλώ, πείτε μας, τι γίνεται με τα hotspot στην Ιταλία και την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Κοινοβούλιο για το αίτημα που μας υπέβαλε να σας ενημερώσουμε για μια γνωμοδότηση που αρχικά είχαμε δημοσιοποιήσει το 2016 για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στα hot spot σε Ελλάδα και Ιταλία πολύ συγκεκριμένη δηλαδή ερώτηση και εκεί θα, σε αυτό το πλαίσιο θα παραμείνω για την απάντησή μου. Την επικαιροποιημένη αυτή έκθεση την ε, δημοσιοποιήσαμε τέλη Φεβρουαρίου πριν λίγες εβδομάδες και μελετήσαμε τον ίδιο αριθμό spot όπως και το 2016 9 τον αριθμό. Υπήρχαν μεν κάποιες αλλαγές στην Ιταλία αλλά ο συνολικός αριθμός παρέμεινε ο ίδιος. Έπρεπε βέβαια να λάβουμε υπόψη για την ανάλυση μας σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες και στις δύο χώρες. Ό,τι αφορά την Ελλάδα μετά ε, την κοινή δήλωση του 16 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ε, άλλαξε η φύση των hot spot ε, αυτών των κέντρων ε, υποδοχής και ταυτοποίησης που δεν ήταν γρήγορη, ε, κέντρα γρήγορης επεξεργασίας αλλά εκεί πλέον διεκπεραιώνονται και οι διαδικασίε υποβολή αίτηση για την παροχή ασύλου. Η προσθήκη τη διάσταση αυτή ε, στα hot spot οδήγησε στην κατάσταση να παραμένουν για πολύ μακρύτερο χρονικό διάστημα εκεί οι άνθρωποι. Πολύ διαφορετικό δηλαδή ε, σε σχέση με το τι αρχικά είχε σχεδιαστεί. Επίσης ένας άλλος παράγοντας για τον οποίο μένουν ε, παρατεταμένες περιόδους στα hot spot οι στην Ελλάδα είναι το ότι δεν υπάρχει ε, μια συνολική ε, προσέγγιση και ένα συνολικό πρόγραμμα με την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, το 16, από το 2016 και μετά άλλαξε η κατάσταση και στην Ιταλία. Αν λάβει κανεί υπόψη το τι έγινε στη Λιβύη με την αρχέτηση ε, και τις ανθρωπιστικές ε, επιχειρήσεις διάσωσης στη Μεσόγειο. Έπεσε σημαντικό αριθμό ε, στην Ιταλία. Δεν έχουμε πρόβλημα υπερπληθισμού, συνοστισμού στα hot spot της Ιταλίας πλέον. Και ένα από τα ε, ζητήματα Είχαμε 21 ε, ζητήματα εντοπίσει το 2016. Στη γνωμοδότηση που τώρα ε, σας παρουσιάζουμε, τα επανεξετάσαμε όλα αυτά τα 21 ζητήματα. Έχουμε βάλει και φανάρια, δηλαδή πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο, για να καταλάβετε τη διαφοροποίηση, την εξέλιξη. Δηλαδή, έχουμε κάποιες τέτοιες εξέλιξεις, δεν είναι όλα ε, ζωφερά. Για να σας δώσω παραδείγματα, στην περισσότερη περίπτωση τα προβλήματα που είχαν να κάνουν με την έλλειψη διεθνούς προστασίας αντιμετωπίζονται αντιμετωπίστησαν στα ελληνικά νησιά με το σύστημα καταγραφής. Το 2019 δεν είχαμε κάποια αναφορά άσκησης ε, περιβολικής βίας κατά τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τώρα, εντοπισμός ευάλωτων ομάδων. Βελτιώθηκε η κατάσταση και στην Ελλάδα και στην Ιταλία στην Ιταλία είχαμε ζητήσει να υπάρξει μεγάλη ενίσχυση των προσπαθειών καταπολέμησης της διακίνησης, παράνομη διακίνηση και με συντονισμό και συνεργασία με την Κομισιόν, ε, τον ΕΑΣΟ, και άλλου κρατικού φορεί βελτιώθηκαν τα πράγματα. Είδαμε επίση πολύ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στην Ιταλία σε ό,τι αφορά τη βία βάση φύλου ή ε, σεξουαλικού προσανατολισμού και πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ε, επίση παιδική προστασία. Υπάρχουν σημεία ε, focal points στην Ελλάδα πλέον γι' αυτό. Επίση, νέοι νόμοι για κυδαιμονία έχουμε και στην Ελλάδα και στην Ιταλία νέου νόμου, Για τα συνόδευτα παιδιά στα Ιταλικά hot spot έχουν γίνει βελτιώσει. και το ίδιο στην Ιταλία. Έχουμε ειδικού χώρου στα περισσότερα hot spot για συνόδευτα παιδιά. Επισκέφτηκα τα hot spot το 2015 και πρέπει να σας πω ότι σήμερα δραματικά έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση προς το καλό ευτυχώς ε, ό,τι αφορά τα παιδιά ιδίω, αλλά υπάρχει και πολλή δρόμος ακόμα αλλά θα σας τα πω στη συνέχεια σε ό,τι αφορά επανεισδοχή και επιστροφές ο Frontex οι συνοδείες ε, από τον ε, οργανισμό αυτό γίνονται, το γραφείο αυτό γίνονται πολύ καλύτερα. Είναι εκπαιδευμένοι συνόδοι πλέον και η ακτοφυλακή, η συνοριοφυλακή εκπαιδεύει του συνόδου αυτού στην Ελλάδα. Επίση έχουμε προγράμματα ε, ελέγχου, υπάρχει παρακολούθηση, ε, σκέπτονται επιθεωρητέ στα hot spot και παρακολουθούν και τις ε, διαδικασίες ε, επιστροφής επανεισδοχής. Άρα βελτιώνονται τα πράγματα, αλλά εξακολουθούν να παραμένουν κενά ε, σε ό,τι αφορά σεβασμό θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα αναφέρω μερικά πράγματα. Σε ό,τι αφορά τους ετούντες άστρους μένουν πέντε μήνες τουλάχιστον, πολύ περισσότερο συνήθως στα νησιά. Και είναι πολύ ε, κακές οι συνθήκες, πολύ κάτω του φυσιολογικού. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα συνοστισμού και σε ό,τι αφορά την παροχή βασικών υπηρεσιών είναι πολύ δυσκή γίνονται οι διαδικασίε, ιδίω ό,τι αφορά του διαγωνισμού. Για να καταλάβετε τι λέω όταν μιλάω για συντονισμό και για ανθρωπιστικέ προκλήσει, μόλι χθε στη ΣΑΜΟ είχαμε 3.949 ανθρώπου σε μια κατάσταση που μπορεί να φιλοξενήσει ουσιαστικά 648 άτομα. Δηλαδή 4.000 άνθρωποι σε μια κατάσταση που μπορεί να φιλοξενήσει 648 κανονικά. Πάω σε άλλα σημεία. Υπάρχουν γνήσιες προσπάθειες σήμερα να ενημερώνται καλύτερα οι ετούντε σα για τι διαδικασίε. Όμω, εξακολουθεί να ισχύει το γεγονό ότι πολλοί ετούντε δεν γνωρίζουν επαρκώ πώ λειτουργούν αυτέ οι διαδικασίε. Υπήρχε ένα πρόβλημα με την παροχή κρατικής, ε, κρατικός χρηματοδοτούμενης ε, νομικής συνδρομής. Ε, στη Γαλλία ένας στη Λέσβο μόνο είναι ο δικηγόρος που χρηματοδοτείται από το κράτος και ο οποίος μάλλον εκεί που έχουμε 4.931 δικηγόρους για 5.000 κάτι, ε, ενώ στοιχείο έναν σε 1.600 τόσους. Έρχομαι στην παιδική προστασία. Διαδικασίες αξιολόγησης της ηλικίας ε, καθυστερούν ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ε, καταφύγει για τα συνόδευτα παιδιά. Δεν είναι ε, επαρκή ούτε ε, πάρα πολύ καλά. Οι συνθήκες κυρίως δηλαδή διαβίωσης δεν είναι καλές εκεί. Βελτιώσεις υπήρχαν. <clears throat> Δηλαδή, εντοπίζουμε του ευάλωτους πιο εύκολα, αλλά υπάρχουν και ένα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν αρκετοί ψυχολόγοι, γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί και διερμηνεί. Και αυτό καθυστερεί πάρα πολύ τι διαδικασίε. Άρα, οι άνθρωποι αυτοί, οι ευάλωτοι, μένουν πολύ μεγάλο διάστημα ε, υπό πολύ άσχημες συνθήκες διαβίωσης ε, σε αυτούς τους χώρους ε. και αυξάνεται η ευαλωτότητά τους τελικά. Η ασφάλεια. Πολύ ένα συνδεδεμένο θέμα. Ξεκολουθούμε να βλέπουμε βία επεισόδια στα hot spots στην Ελλάδα και στην Ιταλία ο συνοσπιτισμός στην Ελλάδα αυξάνει τον κίνδυνο επίσης σεξουαλικής βίας ή βίας βάση φύλου. Σε κάποια ελληνικά hot spot ε, γυναίκες που είναι μόνες τους δεν φιλοξενούνται σε διαφορετικούς χώρους απομονωμένους και οι ε, άνθρωποι που περιπολούν οι αστυνομικοί κυρίως είναι άντρες. αν και γίνεται προσπάθεια να έχουν περισσότερες γυναίκες αστυνομικούς σε αυτούς τους χώρους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση των ατόμων στα hot spot ε, και μιλώ για συγκεκριμένες κοινότητες δεν υπάρχει συμμετοχή επαρκής από την τοπική κοινωνία. Υπάρχουν ε, κενά στην ενημέρωση μεταξύ hot spot πληθυσμού που είναι μέσα στα hot spot και πληθυσμού που τοπικού, εκτός δηλαδή. και πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ τρομερά τα νούμερα. Στο ε, βαθύ της ΣΑΜΟΥ για παράδειγμα, χθε. τοπικός πληθυσμός, ε, οι τοπικοί κάτοικοι 8.000 στον αριθμό και οι μετανάστες που ήταν εκεί 4.201. Και τέλος, ε, πάντως των ανησυχιών που είχαμε εκφράσει, μας ανησυχεί ο βαθμός ε, ε, στον οποίο χρησιμοποιείται η κράτηση ως ε, μέτρο ελέγχου. Στέρηση της ελευθερίας, ε, η δυσανάλογη, είναι προβληματικό θέμα. Και στην Ελλάδα γνωρίζουμε ότι η κράτηση γίνεται ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά του άσυλο που έρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης του ασύλου. Δεν έχουμε να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες συστάσεις στην νομοδότησή μας αγαπητέ πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής και αυτό διότι η επίλυση κατάστασης ε, υπερβαίνει κατά πολύ ε, το δικό μας οργανισμό με τις δικές μας αρμοδιότητες. Τρεις σύντομες παρατηρήσεις και με αυτές θα ολοκληρώσω. είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια μοναπευθυντική θηρίδα όταν κάποιο φτάνει στι ακτέ ενό νησιού. Να υπάρχει ένα σημείο στο hot spot που να αντιμετωπίζονται όλα, να γίνονται όλε οι διαδικασίε. Βέβαια, δείχνει η διαδικασία ότι η επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου στο πλαίσιο του hot spot δημιουργεί ε, μεγάλε προκλήσει ε, σε ό,τι αφορά το ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει οι χαράκτε πολιτικέ να το αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, το δίλημα αυτό, να το λύσουν. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει συνεχή επαγρύπνηση στα hot spot για την ε, προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εμείς θα παραμείνουμε σε εγρήγορση ω οργανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα ε, μόνιμο ε, επίκεντρο και εστίαση σε αυτά τα θέματα. και το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν. Και το τρίτο συμμετοχή της τοπικής κοινότητας, των τοπικών κοινωνίων. Πρέπει να γίνει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να εμπλακούν ε, τα μέλη της τοπικής κοινωνίας, να ακούν, ε, να καταλάβουν περισσότερο, να ε, συμμετέχουν στις αποφάσεις για τον χώρο στον οποίο θα υπάρξουν τα hot spot και το πώς θα λειτουργούν. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Χαίρομαι που τελειώσαμε με αυτό το τελευταίο θέμα. Εγώ προσωπικά γνωρίζω έχω, το θέμα χρειάζεται προσωπικό επιτόπου από τον οργανισμό σας δηλαδή είναι άλλωστε μεγάλα ευρωπαϊκά project και να δείτε τι βελτιώσεις έχουν γίνει, πού παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γνωρίζω ότι έχετε αγωνιστεί ώστε να αποκτήσετε περισσότερη χρηματοδότηση για τις προσπάθειες αυτές γιατί είναι σημαντικό βέβαια τμήμα του έργου σας. Ρωτώ αν επιθυμεί κανείς να λάβει το λόγο για το συγκεκριμένο θέμα. Η Μπάρβαρα Σπινέλη. Σας ευχαριστώ κύριο Φλαχερτή για την παρουσίαση του θέματος. Υπάρχει βέβαια και η κοινή δήλωση, η συμφωνία ας πούμε Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Εάν κατάλαβα καλά από τα όσα είπατε για την αξιολόγηση των hot spot, η αξιολόγηση σας δεν είναι θετική. Για μένα ούτως ή άλλως είναι αρνητική. Αναφερθήκατε σε κάποιες βελτιώσεις, αλλά είπατε και πολλά αρνητικά πράγματα. Κάτι που ρίχνει και κάποιες σκιές σε αυτή τη διστακτική η συγκρατημένη αισιοδοξία. Εγώ θεωρώ ότι η προσέγγιση αυτή έχει αποτύχει. Η προσέγγιση των hot spot. Ίσως να μην συμφωνούμε σε αυτό. Αν όμως δει κανεί και τις πιο πρόσφατες εκθέσεις από τους γιατρούς χωρίς σύνορα για παράδειγμα που έχουν έκθεση για τα hot spots στην Ελλάδα καθώς και άλλοι για την κατάσταση στην Ιταλία. Αυτά προκαλούν, αυτές οι εκθέσεις προκαλούν σημαντικές ανησυχίες ό,τι αφορά την ε, σωματική και ψυχολογική υγεία των ε, προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι κρατούνται στην ουσία στα νησιά αυτά, εφόσον δεν τους επιτρέπεται να τα εγκαταλείψουν. Έχουν δημοσιευτεί και ενδιαφέρουσες ψυχιατρικές μελέτες για την κατάσταση των νέων και των παιδιών. Μιλήσατε για τους νέους. Δεν είμαι βέβαια αν είπατε ότι υπάρχει κάποια πρόοδο. Τα πράγματα όμω είναι ανησυχητικά, διότι πριν από λίγου μήνε είχαμε και ολόκληρη σειρά από αυτοκτονίε ε, νέων ε, σε ελληνικά νησιά και ιδίω στην Μόρια. Έρχομαι στο τελευταίο θέμα. Τα hot spots στην Ιταλία. Δεν είναι εκεί τόσο δραματικά τα νούμερα όσον αφορά δηλαδή την διάρκεια των ορίων των ε, καταβλισμών αυτών, διότι κανείς δεν καταφέρει να φτάσει πλέον στην Ιταλία. Όμως ε, οργανισμοί όπως ο Sea-Watch ε, διαπίστωσαν σημαντικές δυσκολίες για να έρθουν σε επαφή με τους εκπροσώπους τους, ε, του δημοσίου, δηλαδή τα πρόσωπα αυτά τα οποία προσφεύγουν εκεί, για να πληροφορηθούν πώς μπορεί κανείς να καταθέσει αίτηση ασύλου, ας πούμε, πράγματα τα οποία διαφεύγουν εντελώ από όσα προβλέπουν οι διεθνεί συνθήκες. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν και πώς η δουλειά κάνει και πρέπει να κάνει ακόμα ο οργανισμός FRA στον τομέα αυτό. Κορνιλία Έρνστ. Μία ερώτηση. Τα υπόλοιπα τα είπε σωστά η Μπάρβαρα Σινέλη. Θεωρείτε ότι τα hot spot είναι κατάλληλα καταλήματα για ετούντες άσυλο οι οποίοι κάποτε περνούν, ε, διαβιούν μακρό χρόνο εκεί και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγκάζει τις χώρες να εισαγάγουν τον θεσμό των hot spot. Ε, αυτό είναι το περιεχόμενο της ερώτησης μου. Μιχαήλο Φλάχερτη, παρακαλώ αν θέλετε να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ. Πρώτα για την ερώτηση της κυρίας Σπινέλη. Η γνωμοδότηση που αναφέρατε αναφέρεται ειδικά στις εννέα αυτές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, ωστόσο η κατάσταση του μεταναστευτικού και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σχετικά είναι πολύ ευρύτερες. Εγώ θέλησα σήμερα το πρωί να περιορίσω τι παρατηρήσεις μου σε αυτά που είπα. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην κεντρική Μεσόγειο, μας ανησυχεί πάρα πολύ. Ο αριθμός των θανάτων στην θάλασσα. Το, την προηγούμενη χρονιά ήταν κατά μέσον όρο 6 την ημέρα. Και τα πρόσωπα αυτά βεβαίω ποτέ δεν έφτασαν στι ακτέ για να υποστούν οποιαδήποτε μεταχείριση. άρνηση να επιτραπεί στα σκάφη των διασωστών να προσεγγίσουν στα λιμάνια είναι ένα μεγάλο θέμα. Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα των hot spot που έθιξαν και οι δύο ευρωβουλευτές που μίλησαν, η κυρία Σπινέλη και η κυρία Έρνστ. Να υπενθυμίσω πρώτα τι είπα. Είδαμε κάποιε βελτιώσει, παραμένουν όμω πολύ σοβαρά θέματα ανοιχτά. Δεν θέλω δηλαδή καθόλου να σα δείξω ότι δήθεν είμαστε ε, ικανοποιημένοι. Ε, εν μέρη, οι ελλείψει που βλέπουμε οφείλονται στο γεγονό ότι τα spot λειτουργούν με τρόπου που δεν ήταν στον αρχικό σκοπό. Κανονικά θα έπρεπε να μπαίνει κάποιο εκεί και δύο-τρει μέρε να φεύγει. Και εάν γινόταν σεβαστή η χωρητικότητα των hot spot, δεν θα υπήρχαν και όλα αυτά τα ανθρωπιστικά προβλήματα, προβλήματα ανθρωπιστική μεταχείριση, δηλαδή τα οποία σα περιέγραψα. Αυτό που έχουμε τώρα και ιδίω στην Ελλάδα είναι άνθρωποι που είναι στην ουσία αναγκασμένοι να διαβιούν στα νησιά για 5 και 6 μήνε σε πάρα πολύ φορτωμένου καταβλισμού. Και αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Κάτι θα πρέπει να αλλάξει. Όπω για παράδειγμα είπα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταθέσεως και εξετάσεως του αιτήσου ασύλου. Αλλά ακόμη γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει. Ευχαριστώ. Ωραία το είπατε ότι τα hotspot θα διώχναν τους ανθρώπους σε δύο-τρεις ημέρες, θα τους επέτρεπαν να φύγουν δηλαδή, σε δύο-τρεις ημέρες. Ωραία, ε, ε, πολύ ωραία εικόνα που δώσατε. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε ποτέ σε σημείο όπου θα μπορούν, να διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις των ανθρώπων σε δύο-τρεις ημέρες. Ασφαλώς τα ε, hotspot αυτά έφεραν μαζί τους και όλες, όλα αυτά τα προβλήματα που είπατε, τεράστιες καθυστερήσεις κλπ. Χρειάζεται αξιολόγηση ε, των ε, προσεγγίσεων αυτών να γίνουν με κάθε λεπτομέρεια. με κάθε λεπτομέρεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και να ε, αντιλαμβάνουμε ότι είναι μέρο των αρμοδιοτήτων του οργανισμού σα που ελπίζω ότι θα συνεχίσει να δά στοχευμένα. Σα ευχαριστώ. Θα επανέλαβω ναι, αυτό που είπα στην αρχή. Σας ευχαριστώ προσωπικά και ευχαριστώ και το προσωπικό του οργανισμού για όσα έχετε κάνει και ιδίω υπέρ των μελών μας που ήρθαν σε επαφή με τον FRA και συνεργάστηκαν μαζί του. Σα ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Α, εσεί δεν μπορείτε να με ευχαριστήσετε. Δεν θέλω να ακουστεί ότι φεύγω λόγω του ότι είμαι Βρετανός. Αστείευομαι φυσικά. Και εσείς είστε Ιρλανδός, άρα θα παραμείνετε για πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι είναι. Ε, γνωρίζετε ότι προσπαθώ να αλλάξω Εθνικότητα, ε. Επικότητα, διαβατήριο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και είναι πολύ Ρωτώ, Κονίλια, οποιουσδήποτε προσφορές αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος με θέλει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, είναι πολύ καλό αυτό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν 230.000 αιτήσει για ευλαντική ηθαγένεια. Ασφαλώ είναι τεράστια η πρόκληση, οι που αντιμετωπίζεται ω οργανισμό. και πολύ δύσκολο. Όλοι το κατανοούμε αυτό. Και η Σεσίλ θα συμφωνήσει μαζί μου. Δεν με ακούει, αλλά έχουμε και το ψήφισμα για την αφροφοβία για την επόμενη εβδομάδα. Έρχονται λοιπόν και νέε πρωτοβουλίε τις οποίες αναλαμβάνουμε, και αυτές έρχονται και ε, συνδέονται και με το έργο του οργανισμού FRA. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι πολύ τον κύριο Φλάχαρτη. Παρεκάλεσα την Κονίλια ε, Έρνστ να αναλάβει τα ενία της διεύθυνσης για το υπόλοιπο της συνεδριάσεως, γιατί έχω άλλη υποχρέωση. Η Κονέλια λοιπόν θα έρθει για να διευθύνει τη συζήτηση με τους συναδέλφους της Frontex, που όμως δεν έχουν αφηχθεί ακόμη. Άρα, σύντομη διακοπή της τάξης των 10 λεπτών και ευχαριστώ ήδη την Κοσμιλία Ernst που θα προσέλθει για να διευθύνει την συζήτηση. Σε 10 λεπτά. Μην απομακρυνθείτε πολύ. 10 λεπτά διακοπή. Και ευχαριστώ και πάλι Μάικλ

Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 Elhamdülillah.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 Yes, we can open the floor for the colleagues from the group. Λοιπόν, παρακαλώ, οι συνάδελφοι από τις ομάδες, ίσως ε, και το προσωπικό και οι βοηθοί, μήπως μπορούν να... Θέλει κανείς το λόγο. Ας περιμένουμε.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

Okay, I think, uh, I think we can start our last um, panel in... Λοιπόν, τελευταίο μας θέμα. Συμβουλευτικό φόρουμ ε, Frontex για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το επόμενο θέμα. Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης 2018 από την κυρία Βαγεστέρο που είναι πρόεδρος ε, του φόρουμ και από τον κύριο Κέσλερ. που είναι ανώτατος υπάλληλο, Είναι και οι δύο ε, συμπρόεδροι του Συμβουλευτικού Φόρουμ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Εμεί ως ομάδα τη αριστερά ε, προτείναμε να προσκληθείτε. Συνεργαζόμεθα και χαιρόμαστε πολύ για τη συνεργασία μα και για την παρουσία σα. Οπότε, η κυρία Βαγεστέρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή που μας ε, προσκαλέσατε εκ νέου για να σας υποβάλουμε την εργασία μας κατά τη διάρκεια του 2018. Άλλη μια ε, χρονιά αλλαγών και πιέσεων για να εκτελέσει την αποστολή της Ιφράντεξ και από πλευράς της αρμοδιότητάς της, της ευθύνης της για τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ολοκλήρωση του, των συμφωνιών με τις χώρες των, Δατικών, των Δυτικών Βαλκανίων και η προώθηση των συζητήσεων που ξέρετε για την έγκριση του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή 2.0 καθώς και η έκρηση του κανονισμού ETIAS ε, είναι μερικέ από τι προκλήσει που αντιμετωπίσαμε πέρυσι. Και ε, φέτο όμω θα έχουμε και άλλε προκλήσει. Αλλάζει η κατάσταση στο Συμβουλευτικό Φόρουμ. Έγινε μια εξωτερική αξιολόγηση τη εργασία μα που θα ολοκληρωθεί και ελπίζουμε να εμπνεύσει το μέλλον των εργασιών μας και θα μας στηρίξει και θα μας συμβουλεύσει για την ε, σύνθεση του φόρου μας που θα αλλάξει φέτος. Η συμμετοχή σας στη δημιουργία και τη λειτουργία του φόρου μας και της εργασίας μας θα είναι κλειδί σε αυτή την αξιολόγηση και θα συμμετάσχετε επαρκώς σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα τα θέματά μας. Η έκθεσή μας σας έχει διανεμηθεί. Ελπίζω να τη διαβάσατε. Παρουσιάζει σωστά την κατάσταση, νομίζω ότι είναι εύγλωτη, αλλά φυσικά να συμμετάσχουμε στη συζήτηση για να υπάρξει δούνε και λαβίν. Να υπογραμμίσουμε μερικά από τα βασικά στοιχεία της δουλειάς μας πέρυσι. Πρώτον, η συνεχόμενη και αυξανόμενη ε, δουλειά μαζί με τις χώρες. Έχουμε ενισχύσει τη δουλειά των ε, υπευθύνων σύνδεσης με τις χώρες. Επισκεφθήκαμε τα Δυτικά Βαλκάνια για να συζητήσουμε επί τόπου την κατάσταση. Έχουμε κάνει και διάφορες συζητήσεις με τους υπευθύνους σύνδεσης και με την υπηρεσία στήριξης που έχουμε δημιουργήσει στον Frontex για να τους βοηθάει και θα κάνει ο οργανισμός μας, ο φορέας μας, μια γενικότερη συζήτηση εστιάζοντας στο ρόλο αυτών των υπευθυνών σύνδεσης για την πρόθεση των ε, κανόνων για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είχαμε και πέρυσι μια μελέτη που απαιτέλεσε τη βάση για μια σύσταση για τις επαφές μας με τρίτες χώρες και συμπίπτει με την έναρξη των ε, επιχειρήσεών μας στα Δυτικά Βαλκάνια. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η εκπόνηση αυτών των συστάσεων και θα αποσταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο προσεχώς. Δεύτερο τμήμα του οργανισμού μας που ε, απασχολεί το φορέα μας είναι το θέμα των απάτριδων άτομα χωρίς ε, ηθαγένεια είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια συγγνώμη Ε, μισό εκατομμύριο εξ αυτών είναι στην Ευρώπη. Είναι δύσκολο να εντοπιστούν τα άτομα αυτά. Αναγνωρίζουμε ότι πολλοί από αυτούς που φτάνουν στην Ευρώπη είναι από χώρε όπου υπάρχουν πληθυσμοί απάτριδων, όπως είναι η Συρία, το Ιράκ, η Ερυθρέα ή το Αφγανιστάν, όπου υπάρχουν ε, πολλά άτομα χωρίς ηθαγένεια. Στην ε, σύστασή μας λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να συμβάλλει ο οργανισμός μας, ο Frontex, στην αντιμετώπιση του φαινομένου μέσω του ρόλου που έχει στα σύνορα αλλά και δημιουργούντας προδιαγραφές και πρακτικές για τον καλύτερο εντοπισμό και καταγραφή αυτού του πληθυσμού. Πιστεύουμε ότι έτσι θα λάβουν περισσότερη προστασία και θα επιτρέψει στην Frontex να επιτελέσει το έργο του συλλογή ακριβών στοιχείων, δηλαδή με ακρίβεια στοιχείων, και καλύτερη προπαρασκευή της αντιμετώπισης μέσω των λειτουργιών μας και μέσω της στήριξης που δίνουμε στα κράτη-μέλη. Τρίτο σημείο. Προστασία των παιδιών και θέματα φύλου. Έχουμε ασχοληθεί πολύ με τα θέματα αυτά στο παρελθόν και κατά τη διάρκεια του 2018 συνεχίσαμε αυτή την ε, εστίαση στα θέματα αυτά. Και εδώ χαιρετίζω τις προσπάθειες της Frontex που, που εφήρμοσε μία από τις ε, συστάσεις μας. Έχουν και λεπτομεριακά στοιχεία για την ηλικία και το φύλλο. Αυτό έχει βελτιώσει τη δυνατότητα που έχει η Frontex να προετοιμαστεί και να ε, εφαρμόσει τις πολιτικές της για να βοηθήσει τις αντίστοιχες ομάδες και αυτό σχετίζεται με καλύτερη καταγραφή όπως και με το προηγούμενο θέμα του ποιοι φτάνουν, πόσοι φτάνουν και και με ποιους χρειάζεται να ασχοληθούμε. Και τέταρτο και τελευταίο. Το θέμα της κατάρτισης. Ε, και η κατάρτιση επειδή επεκτείνεται συνεχώς η Frontex και σε τρίτες χώρες ε, γίνεται όλο και πιο σημαντική. Επεκτηνόμεθα και σε περιοχές όπου υπάρχουν υψηλότεροι κίνδυνοι όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Βεβαίως το προσωπικό μας ε, είναι ιδιαίτερα ευσυνείδητο και κάνουν αυτά που είχαμε αποφασίσει, έχουν συμβάλει στις προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή και αυτή τη στιγμή έχουμε μια διαδικασία εντοπισμού και καταγραφής μαζί με την Frontex για να καταλάβουμε καλύτερα με τι θέματα ασχολείται τώρα η κατάρτισή μας για να δώσουμε και καλύτερες συμβουλές όσο αυτός ο τομέας αρμοδιοτήτων της ε, Frontex επεκτείνεται. Και τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Στέφαν. Είμαστε το σύνηθες ντουέτο. Το ένα μέρος η Μάρτα, το άλλο εγώ. Θα προσθέσω τέσσερα ε, σημεία στα όσα είπε. Πρώτο, Έχουμε ζητήσει έξτρα χρηματοδότηση για ορισμένα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσα στα πλαίσια ε, ε, επιχειρήσεων με πλήονες φορείς. Υπάρχουν και άλλοι φορείς λοιπόν οι οποίοι εμπλέκονται στις ε, αποστολές μας και για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαμε δυσκολία να ορίσουμε ποιος είναι υπόλογος για ποιο πράγμα. Δεν είναι εύκολη υπόθεση ούτε εύκολο το ε, αντικείμενο. Έχουμε εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κάνουν τη σχετική ανάλυση. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε επί των συστάσεων. Πάντως από τις πιο σημαντικές εκβάσεις της συνάντησης ε, των εμπειρογνωμόνων ήταν να τονιστεί η ανάγκη της γνώσης και αφενός η Frontex να αφιερωθεί στη συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών, δηλαδή δεν μπορούν απλώς να περιμένουν με σταυρωμένα χέρια, θα πρέπει να δράσουν ενεργά ώστε να εμπλακούν στην θέσπιση μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι συλλέγεται, συλλέγονται σχετικές πληροφορίες. Από την άλλη μεριά, σημαντικός ο, και κύριος ο ρόλος του αξιωματούχου για τα, για τα θεμελιώδη δικαιώματα που συμβάλλει στην ε, δημιουργία της σχετικής αυτής γνώσης. Μίλησα για το Fundamental Rights Officer η συνεργασία με τον αξιωματούχο αυτό στην Frontex έχει τεράστια σημασία για μας. Ακόμα περισσότερο που βασίζεται ο οργανισμός στην ανεξάρτητη, στον ανεξάρτητο αυτό αξιωματούχο ή ανεξάρτητο γραφείο για τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα. Και ευχαριστούμε και για την εμπλοκή της δικής σας επιτροπής για να υπάρξει η αναγκαία στελέχωση του γραφείου. Θυμίζω τη γνωμοδότησή σας για την απαλλαγή του Frontex για το έτος 2017, όπου σωστά περιλαμβάνεται το εξής. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της συνολικής αύξηση προσωπικού του οργανισμού, εξακολουθεί το γραφείο να στερείται της αναγκαίας στελέχωσης που δυσχεραίνει το έργο του. Πόσο καλύτερα να το λέγαμε και εμείς οι ίδιοι. Μια μικρή αύξηση των μελών του προσωπικού υπήρξε για το Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, διότι προσελήφθη ένα πρόσωπο το 2018 σε θέση βοηθού όμως ο τρέχον διαγωνισμός δεν επιτρέπει να αναμένουμε να ε, προσληφθεί επαρκές προσωπικό για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και ακόμα χειρότερα δεν υπάρχει δομή που να επιτρέπει να ασκούνται από άλλους τα καθήκοντα του γραφείου. Έχουμε δηλαδή το πρόβλημα ότι ο αξιωματούχος θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι σε παρατεταμένη άδεια ασθενείας έχουν βάλει μια προσωρινή αντικατάσταση ένα πρόσωπο θηλυκού γενούς το οποίο βέβαια ε, απαράχθηκε από τα καθήκοντά της το ε, προσωπικό γραφείο και έχει αναλάβει τα καθήκοντα του αξιωματούχου θεμελιώδων δικαιωμάτων. Πάντως, για το λόγο αυτό, διακυβεύεται τώρα η ανεξαρτησία του αξιωματούχου θεμελιών δικαιωμάτων. Δεν έχει γίνει και αξιολόγηση του μηχανισμού υποβολής παραπώνων. Εμείς κάναμε, ε, ε, έχουμε υποβάλει σχόλια για τον μηχανισμό υποβολής παραπώνων και χαιρόμαστε για τις προσπάθειες που κάνει ο αξιωματούχος θεμελιών δικαιωμάτων και έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση. Αλλά δεν είχε γίνει αξιολόγηση εκ των προτέρων. Δεν είμαστε βέβαιοι λοιπόν εάν οι διάφορες ανεπάρκειες που είχαμε διαπιστώσει έχουν αντιμετωπιστεί και θεραπευτεί με τη νέα ρύθμιση. Και μας ανησυχεί ακόμα η προσβασιμότητα του μηχανισμού υποβολής παραπώνων από τα πρόσωπα που θέλουν να υποβάλουν παράπονα. Και τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην αναθεώρηση της στρατηγικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα του Frontex Τη οποία τελευταία εκδοχή είναι χρονολογείται το 2011. Από τότε όμως ο κόσμος έχει αλλάξει αρκετά, ιδίω στο πεδίο αρμοδιότητας του Frontex. Όμως εξακολουθούμε να έχουμε ακόμα την παλαιά στρατηγική και παρόλες τι επανειλημμένες εκκλήσει μας για νέα αξιολόγηση, για νέα στρατηγική, το πρόβλημα ακόμη δεν έχει λυθεί. Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι να ε, βοηθήσουμε στο έργο αυτό και κατά τη γνώμη μας ο τελικός στόχος θα πρέπει να είναι η στρατηγική θεμελιδών δικαιωμάτων να απηχεί την αύξηση των του ε, οργανισμού Frontex. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είμαστε βεβαίως στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Thank you Uh, Η Προεδρεύουσα Κορνίλια Έρνστ, σας ευχαριστώ πολύ για τις σημαντικές παρεμβάσεις που είχαν και κριτικό χαρακτήρα. Επιτρέψτε μου να δώσω πρώτα το λόγο στην, στις μου, προκειμένου στην Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ, Κόνη. Κυρίως Θέλω να σε ευχαριστήσω και για την πρωτοβουλία. Να ευχαριστήσω και τους κυρίους ε, από τη Frontex για το έγγραφο, την κυρία Μπαλιστέρη και τον κύριο Κέσλερ. Έχω δύο ερωτήσεις, τις οποίες θα ήθελα να θέσω. Στη δουλειά μου ως εισηγητρία για το χάρτη των δικαιωμάτων διαπίστωσα ότι η Frontex έχει έναν αρκετά καλό οργανωμένο μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε αντίθεση με άλλους οργανισμούς. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι ορισμένα στοιχεία καθιστούν συχνά αναποτελεσματικούς αυτούς τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και αυτό το επιβεβαιώνει και η δική σας έκθεση είτε σε ό,τι αφορά τους πόρους είτε σε ό,τι αφορά ιδίως την ανεξαρτησία ε, του ειδικού ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σελίδα 20 συγκεκριμένα. Γίνεται λόγος για τον αναπληρωτή διευθυντή ο οποίος επελέγει στο πλαίσιο της ασταλιστικής εξουσίας ε, της Frontex, αλλά ήταν μια κατάφορη περίπτωση παραβίασης ε, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων. Και στην έκθεσή σας τα λέτε αυτά και θα ήθελα να ακούσω αν ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex αντέδρασε επ' αυτού του περιστατικού. Διότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της ανεξαρτησίας. Επίσης θα ήθελα να μάθω τι γίνεται με το μηχανισμό υποβολής καταγγελιών. Ο κύριος Κέσλερ νομίζω είπε πως υπάρχει βαθιά ανησυχία. Δεδομένων των δυσκολιών πρόσβασης στο μηχανισμό υποβολής καταγγελιών. Επομένως, θα ήθελα να μου πείτε τα εκτελεστικά στελέχη της Frontex πώς έχουν αντιδράσει απέναντι και σε αυτό το ζήτημα. Έρχομαι σε ένα άλλο. Θέμα του όλο και αυξανόμενου ρόλου της Frontex στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό διότι η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδόν 100% βασίζεται στην εξωτερήκευση της ε, πολιτικής ασύλου και στην πολιτική των λίγο πολύ καταναγκαστικών ε, επαναπατρισμών. Ο ρόλος της Frontex αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι θα ενισχυθεί ιδιαίτερα. και νομίζω ότι θα δούμε μια συγχώνευση μεταξύ εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, δηλαδή των πολιτικών που είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και των πολιτικών των εσωτερικών πολιτικών Άρα εσωτερικέ πολιτικέ, ε, όπω οι πολιτικέ ε, για τα εσωτερικά αισθήματα και τη δικαιοσύνη, θα αναμειγνύονται πλέον με τα θέματα εξωτερική πολιτική. Αυτό με ανησυχεί. Θα ήθελα να ακούσω και τη δική σα άποψη. Γιατί η Frontex θα μπορούσε να δραστηριοποιείται από εδώ και πέρα πολύ περισσότερο και σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή θα έχει ρόλο και σε τρίτες χώρες, τρίτες απέναντι στην Ένωση χώρες. βλέπουμε εκτός ε, του διεθνούς δικαίου να γίνονται πολλές επαναπροωθήσεις. Ε, κυρία Πρόεδρος, ε, θα ήθελα να παρακαλέσω την Κομισιόν να πάρει το λόγο εφόσον έχει να σχολιάσει κάτι. Φαίνεται ότι δεν έχετε κάτι να σχολιάσετε από την υπετέρμαστε για τους πρόσφυγες, ούτε κι εσείς. Ουδέν σχόλιον. Καλώς. Τότε εγώ έχω ερωτήσεις, αν μου επιτρέπετε, και θα τα πω στα γερμανικά. Για σας πρώτα κύριε Μπαλεστέρο. Μιλήσατε για τους απάτριδες και είπατε ότι είναι σημαντικό πρόβλημα, μιλήσατε και για νούμερα κατ' εκτίμηση. Ίσως μπορείτε να μας πείτε πού νομίζετε ότι εντοπίζεται η ανάγκη να αναλυφθεί η δράση, δηλαδή τι θα πρέπει να γίνει πρώτα-πρώτα, ώστε να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση των απατρίδων Είπατε ότι θέλετε να επεξεργαστείτε κοινά πρότυπα. Προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί αυτό. Και δεύτερο, μιλήσατε για προστασία παιδιών και για θέματα ισότητας φύλων. Πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Ένα μέγα θέμα είναι βέβαια εν προκειμένου και οι έγκυοι γυναίκες. Ε, το έχετε αυτό ας πούμε ε, μέσα στη στόχευσή σας. Έγκυοι γυναίκες που βέβαια βρίσκονται σε, ιδιαίτερα, σε πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Και τα ζητήματα ε, εκπαίδευση που βρίσκεται να είναι οι μεγαλύτερε ελλείψει. Για τον κύριο Κέσλερ ήδη ερώτησε η συνάδελφός μου Σπινέλη. Αν θέλετε μπορούμε να αρκεστούμε σε αυτά τα ερωτήματα. Καλά λοιπόν. Να σας δώσω το λόγο και αν θέλετε μπορείτε να αποφασίσετε ε, ποιος θα απαντήσει πρώτος, ο κύριος Κέσλερ ή η κυρία Μπαλιστέρα. Ας αρχίσουμε λοιπόν ανάποδα τώρα, θα, πρώτος εγώ και μετά να ακολουθήσει η κυρια ας αρχισουμε λοιπον Νομίζω απήντησε ήδη στην κυρία Σπινέλη. Με τον εκτελεστικό διευθυντή στις συζητήσεις και με το management έχουμε θέσει το θέμα της ανεξαρτησίας του αξιωματούχου ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και που έχει αντικασταθεί από μέλος τώρα του ε, Διοικητικού Συμβουλίου. Ως τώρα η απάντηση πάντως ήταν ότι δεν βλέπουν να υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν με εξέπληξε πολύ. Το επιχείρημα που προέβαλαν ήταν ότι είναι προσωρινή η κατάληψη θέση αυτής. Και εφόσον απαλλάσσεται από τα καθήκοντά της ως μέλους ε, ε, του Συμβουλίου, δεν θα υπάρχει ε, εξάρτηση. Μην πυροβολεί τον πιανίστα θα πω εγώ. Σας αναφέρω απρός τι μας απήντησαν. Για το μηχανισμό υποβολής παραπώνων είπα ότι βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης ή επανεξέταση καλύτερα. Νομίζω ότι έχει βελτιωθεί επί τα βελτίω. Έχει βελτιωθεί προς το καλύτερο δηλαδή. Και σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα στο μηχανισμό υποβολή παραπώνων, αυτό μας ανισχύει βεβαίω. Μου είπε η γερμανική συνοριοφυλακή, για παράδειγμα, ότι έχει κάτι μακροσκελέστατα έντυπα όπου μπορούν ε, να γράφουν τα παράπονά τους, αλλά δεν μου απάντησαν αρκετά. Στο ε, ερώτημά μου, λέτε στον κόσμο ότι μπορεί να πάρει το έντυπο και να ε, υποβάλει τα παράπονα του ή περιμένετε να σας το ζητήσει κάποιος. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί για τον αυξανόμενο ρόλο του Frontex. Κυρία Σπινέλη, νομίζω ότι σχολιάσατε εσείς ίδια το νέο έγγραφο EBCG με την επέκταση του ρόλου, επέκταση των αρμοδιοτήτων ε, του νέου ρόλου δηλαδή των ε, συνοριοφυλάκων και αυτοφυλάκων και για τη δυνατότητα συνεργασίας με τρίτες χώρες. Αν κατάλαβα καλά, ο εισηγητής του νέου κανονισμού θα υποβάλει στην Επιτροπή τα πρώτα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο τότε καλύτερα να τεθούν οι ερωτήσεις γιατί ως συμβουλευτικός φορέας δεν μπορούμε να ε, σχολιάσουμε ακόμα. Θα μπορούσα ε, προσωπικά βέβαια να απαντήσω πολύ μακροσκελέστερα. Όχι όμως για το συμβουλευτικό φόρουμ. Εκεί πρέπει να ε, αυτοπεριοριστώ. Η κυρία Μπαλεστέρο. Λοιπόν, για τους απάτριδες κάτι που καταλάβαμε κάτι διάρκεια της χρονιάς είναι ότι δεν ε, υπάρχει και γνώση του θέματος. Δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση για το θέμα των απάτριδων. Ένα σημαντικό καθήκον που η Frontex ε, μπορεί να βοηθήσει είναι ε, να υπάρξει ευαισθητοποίηση, να μην είναι πια αόρατα τα άτομα αυτά. Να γνωρίζουμε ότι όταν έχουμε τέτοια άτομα στα σύνορα <clears throat> μπορεί να υπάρχει αυτό το πρόβλημα και ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν σωστά. Οπότε κυρίως ε, εστιάζουμε στην, ε, στα καθήκοντα και το ρόλο που μπορεί να παίξει η Frontex. Αυτή λοιπόν πρώτα απ' όλα η καταγραφή, η ευαισθητοποίηση, σωστή κατάρτιση ούτως ώστε όλοι οι ε, <clears throat> υπάλληλοι στα σύνορα να γνωρίζουν ποιο είναι το πρόβλημα, να γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση στη Συρία που μπορεί να καταλήξει με άτομα ε, να γίνονται απάτριδες, πώς ε, <clears throat> οι νόμοι ε, στις εθνικές νομοθεσίες προβλέπουν την μεταβίβαση της υπηκότητας από τη μητέρα στα παιδιά, τι μπορεί να προκύψει και αν κάποια παιδιά γεννηθούν καθοδόν ή αν υπάρχουν περιπτώσεις γονέων που δεν μπορούν να ε, περάσουν την υπηκότητά τους στα παιδιά τους πρέπει γρήγορα ε, να εντοπίζονται αυτές οι περιπτώσεις και να υπάρχουν οι κατάλληλες διαδικασίες ούτως ώστε οι αρμόδιες αρχές να καθορίσουν το καθεστώς του ατόμου που θα μπορούσαν ενδεχομένω ε, χωρίς υπηκότητα Όλα αυτά είναι πολύ βασικά. Στη δουλειά της Frontex. Ούτως ώστε <clears throat> να γίνει κάθε προσπάθεια για να αποφευθεί παραταταμένη περίοδος κράτησης που μπορεί να αποφευθεί Αν ξέρεις από τη στιγμή ε, ποια είναι η κατάσταση, να εντοπίσει από τη στιγμή άφηξής του, αν γίνει σωστά <clears throat> η εξακρίβωση των στοιχείων του, μπορεί να βοηθήσει την όλη διαδικασία. Ε, <clears throat> γιατί αν έχει ένα άτομο υποκράτηση, το οποίο δεν μπορεί να επιστραφεί κάπου, γιατί η χώρο που θα ήθελε να επιστραφεί δεν τον αποδέχεται για λόγους πικότητας, όλα αυτά θα μπορούσαν να δουλεύουν καλύτερα. Μέσω περισσότερης ευαισθητοποίησης, καταγραφής, εξακρίβωσης και έχουμε κάνει συγκεκριμένες συστάσεις. Φυσικά και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να κάνουμε για τους απάτριδες, <clears throat> αλλά αυτά τα σημεία έχουν να κάνουν με την εργασία της Frontex. Θέματα φύλου, προστασία των παιδιών και εδώ. Το θέμα είναι οι αρμοδιότητες της Frontex. Όπως είπε ο συνάδελφος, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για τις απόψεις ε, του υπάτου εκπροσώπου για τους πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών για το θέμα αυτό, αλλά θέλουμε να ασχολούμαστε με τον εντοπισμό αυτών των ε, ατόμων μόλις φτάνουν στα σύνορα. Το προσωπικό στα σύνορα είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι τα πρώτα άτομα με τα οποία έρχονται σε επαφή αυτά τα άτομα. Πρέπει λοιπόν να είναι σωστά καταρτισμένοι, να έχουν τη σωστή ενημέρωση για να εντοπίσουν τα ευάλωτα άτομα και τις ε, εγγύους. Και έχουμε προτείνει στην Frontex τι πρέπει να κάνει και ο αρμόδιος για τα, ανθρώπινα, για τα θεμελιώδη δικαιώματα έχει την αναγκαία πληροφόρηση για να ε, γίνονται οι σωστές διαδικασίες να καθοριστεί εάν ένα άτομο είναι έγκυος και να δράσουμε γρήγορα. Νομίζω ότι εκεί θα μπορούσε να βοηθήσουμε να παίξει καλύτερα το ρόλο της ε, η Frontex. Ευχαριστώ πολύ για την ε, συμβολή σας. Θέλετε να πείτε κάτι ακόμη. Κάτι είχατε πει για ένα τρίτο σημείο για την ε, Κάτι είπατε για την κατάρτιση, αλλά δεν θυμάμαι τι είπατε. Τι ρωτήσατε. Πού υπάρχουν σημαντικές, σημαντικές αδυναμίες στην κατάρτιση. είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα. Να υπάρχει συνέχεια η Φράντεξ καταρτίζει το προσωπικό της για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους συνοριοφύλακες, αλλά έχουμε όλο και αντικατάσταση του προσωπικού. Αλλάζουν πολύ γρήγορα και δεν υπάρχει ε, συνέχεια. Δεν είμαστε σίγουροι ότι ο κάθε συνοροφύλακας που συμμετέχει σε μία επιχείρηση έχει λάβει την κατάλληλη κατάρτιση. Ορισμένες φορές υπάρχει θέμα γλώσσας. δεν ξέρουν όλοι αγγλικά. Οπότε υπάρχουν προβλήματα επικοινωνία. Δεν ξέρω αν έχει να πει τίποτα άλλο. Ναι. Ναι, θέλουμε να εντοπίσουμε καλύτερα τις ανάγκες ούτω ώστε να καταρτιστούν σωστά όλοι οι συνοριοφύλακες και προτείνουμε στη Frontex να υπάρχουν οι σωστοί μηχανισμοί ε, να ελέγχεται ότι οποιοδήποτε δουλεύει σε μια επιχείρηση, σε ένα κράτο μέλος ε, ή τώρα και σε μια τρίτη χώρα ε, προσεχώς δηλαδή, θα έχει λάβει ενημέρωση για τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, απάτριδων, ε, δικαιωμάτων των παιδιών, να είναι πλήρως καταρτισμένος. Και αυτή η διαδικασία καταγραφής που έχουμε θα μας βοηθήσει να ξέρουμε και τι κατάρτιση μπορούμε να προτείνουμε τα επόμενα χρόνια η Πρόεδρος. Βεβαίως πολλά έχουμε να κάνουμε. Άκουσα και τις επικρίσεις, άκουσα και τις συστάσεις, πολλά έχουμε μπροστά μας. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να επιτύχουμε περισσότερα τα επόμενα χρόνια. Και σας ευχαριστώ και για την τεκμηρίωση. Ευχαριστώ που είστε εδώ και τώρα καλή όρεξη.